πληρωμών 38,9 εκατομμύρια ευρώ και το 75% έχει εκτελεστεί. Πρόκειται λοιπόν για προγράμματα τα οποία έχουν ως στόχο την πρόληψη τόσο της τρομοκρατίας όσο και της εγκληματικότητας. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Παριά που απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις. Πάμε στην επόμενη κοινή συζήτηση σχετικά με τον Frontex. Είναι τα σημεία 4, 5 και 6, γιατί είπαμε να μην μιλήσουμε για το 7, αναμένοντας περισσότερες πληροφορίες από Κομισιόν και Συμβούλιο. Καταρχήν, να καλέσω τον εκτελεστικό διευθυντή, την εκτελεστική διευθύντρια του ε, της Frontex την κυρία Λάιτινεν, η οποία θα μας μιλήσει για τους τομείς προτεραιότητας της Frontex για το 2010. Διαδικαστικά ο κύριος Μπουσουτήλ. Επιτρέψτε μου να πω το εξής. Εδώ μιλάει για την παρουσίαση του προγράμματος του 2010. Θα ήθελα η κυρία Λάιτινεν όμως να κάνει και μια αναφορά σχετικά με τα πεπραγμένα του 2009 γιατί θα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να ξέρουμε τι έκανε ο οργανισμός πέρσι όχι μόνο τη σχεδιάζει για φέτος, επίσης να πω ότι μέχρι τώρα δεν λάβαμε αντίγραφο του προγράμματος εργασίας, οπότε δεν διαβάσαμε τίποτα πριν από τη συνάντηση αυτή στο μέλλον. Ίσως θα έπρεπε να παίρνουμε τα έγγραφα αυτά εκ των προτέρων. Ευχαριστώ κύριε Μπουσουτήλ. Συμφωνώ 100% με αυτό που είπατε στο τέλος. Και αυτό αφορά οποιαδήποτε πληροφορία. Α, ε, ο κύριος Λάιτινεν, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Ο κύριος Λάιτινεν θα παρουσιάσει το θέμα του, αναφερόμενος και σε αυτό το αίτημα του κυρίου Μπουσουτήλ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και όλα τα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, όπως και όλους τους παρευρισκομένους. Εύχομαι κάθε, πολλές επιτυχίες το 2010 και Πολύ ε, χαίρομαι που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να έρθω και να παρουσιάσω το πρόγραμμα εργασίας του 2010 στην Επιτροπή σας. Ένας λόγος για τον οποίο δεν υπέβαλα το ίδιο το έγγραφο είναι ότι ακόμα δεν έχει επισήμως ε, εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτό θα γίνει στις 2 Φεβρουαρίου για διαδικαστικούς και δημοσιονομικούς λόγους ε, γιατί δηλαδή επίσημα δεν έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο το πρόγραμμα εργασιών του 2010. Δεν προβλέπονται αλλαγές, απλώς ε, έτσι έχει το χρονοδιάγραμμα. Χώρισα την παρουσίασή μου σε 12 κεφάλαια θα προσπαθήσω να είμαι πολύ εστιασμένος, δεν θα ε, ε, τα αναλύσω όλα με τον ίδιο τρόπο, θα περιοριστώ στα πιο ενδιαφέροντα και σε ένα σημείο θα επικεντρωθώ στα αποτελέσματα του 2009. Και ελπίζω ότι θα καλυφθεί έτσι ο κύριος Μπουσουτήλ. Θα πω αρκετά πράγματα. Η γενική έκθεση πεπραγμένων αργότερα θα κυκλοφορήσει. Τώρα, για το 2010 πρέπει να πω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά για τη Frontex, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα επιτάπητος, αρχίζοντας με τη συνθήκη της Λισαβόνα το πρόγραμμα της Στοκχόλμης και το γεγονός ότι πρόκειται και ο κανονισμός του οργανισμού να τροποποιηθεί μετά από πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτό αποτελεί πρόκληση βεβαίως και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα συμμετάσχει επίσης στα εγχειρήματα αυτά. Είναι πολλές οι προκλήσεις που πρόσφατα είδαμε και που δημιουργούν ε, με τη σειρά τους προκλήσεις στη Frontex. Τώρα, οι στόχοι και οι αξίες της Frontex έχουμε τέσσερις στόχους. Έχουμε την ε, ε, παρακολούθηση που πρέπει να βελτιωθεί, θα πρέπει να υπάρχουν αντιδράσεις, θα πρέπει να υπάρχει διαλειτουργικότητα και απόδοση. Η απόδοση δηλαδή ε, είναι το γενικότερο. Και σε ό,τι αφορά τις αξίες, ε, ανθρωπισμός είναι το υπαριθμόν ένα, ανοιχτή επικοινωνία, επαγγελματισμός, και αξιοπιστία. Εμπιστολές είναι οι αξίες που διέπουν τη στρατηγική, το ετήσιο πρόγραμμα και τις επιχειρησιακές στρατηγικές. Δύο λόγια τώρα για την κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να παρουσιάσω όλη την εικόνα για το, από το 2009, γιατί τα στοιχεία και οι αναλύσεις από το τελευταίο τρίμηνο δεν είναι ακόμα έτοιμα. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση από την πρώτη μέχρι, από το πρώτο μέχρι το τέλος του τρίτου τριμήνου. Ε, παράνομες είσοδοι στα σύνορα και απορρίψει εισόδου ήταν 165.700, μείωση κατά 22%. Στατιστικά σημαντική μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008, αυτό το μείον 22%. 22% μείωση. Τώρα, ε, πώς επιμερίζονται αυτά τα περιστατικά. Είναι πολύ χρήσιμο να έχουμε υπόψη μας ότι κάθε δεύτερο περιστατικό, όταν πρόκειται δηλαδή για παράνομες εισόδου και αρνήσεις εισόδου, ε, στα χερσαία σύνορα λαμβάνει η χώρα κάθε δεύτερο περιστατικό και τα υπόλοιπα μοιράζονται. Θαλάσσια σύνορα 24% και ε, αερία 26%. Κάθε δεύτερη λοιπόν παράνομη είσοδος ή απόρριψη ε, λαμβάνει η χώρα στα χερσαία σύνορα. Τώρα, ας δούμε τους άλλους τομείς, ε, όπου, δηλαδή ε, λαμβανει χωρα στα χερσαια συνορα παράνομη παραμονή, 250.000 περίπου, ε, το πρώτο εννεάμινο, πάλι έχουμε πολύ σημαντική μείωση, μείον 30%. Ε, παραποιημένα ε, έγγραφα, περίπου 10.000 περιστατικά. Αυτό το ποσοστό, αυτός ο αριθμός δεν είναι πολύ μεγάλος. Δουλεύουμε σκληρά, γιατί ξέρουμε ότι τα παραποιημένα έγγραφα και η χρήση τους είναι ο πιο συνήθις τρόπος ε, λειτουργίας και τρόπος, τρόπος λειτουργίας των παρανόμων μεταναστών. Θέλουμε να ε, αυξήσουμε μπορέσαμε να αυξήσουμε σε αυτό το χρονικό διάστημα τον εντοπισμό των διακινητών ε, κατά, έχουμε καλύτερα ποσοστά κατά 15% συγκεκριμένα. Το ίδιο ισχύει και για τους ετούντες άσυλο. Οι ετούντες άσυλο ε, δεν αποτελούν απειλή, αυτή καθ' αυτή. εμάς μας ενδιαφέρουν όμως οι ψεύδο αιτήσει ασύλου και αυτό θα το δούμε και αργότερα. Ας δούμε τώρα πώς κατανέμονται γεωγραφικά όλα αυτά. Ε, χρησιμοποιούμε αυτές τις ε, φούσκες όπου είναι πράσινες οι φούσκες, αυτό είναι καλό. Όπου η φούσκα είναι πορτοκαλί ε, είναι τα πράγματα αμετάβλητα και όπου είναι κόκκινη η φούσκα εκεί τα νέα είναι άσχημα. Μπορούμε να πούμε ότι στα Κανάρια νησιά παρουσιάζεται δραστική μείωση σε σχέση με το 2008. Τα στοιχεία το 2009 συνολικά θα είναι λιγότερο από 3.000, ενώ πριν από δύο χρόνια είχαμε 30.000. Οπότε έχουμε λιγότερο από 10% τώρα ε, τέτοιου είδους περιστατικά στα Κανάρια νησιά. Ιταλία, Μάλτα, Κεντρική Μεσόγειος δηλαδή, μετά το Μάιο, μετά το Μάιο ε, μπορέσαμε να κλείσουμε αυτή την οδό διακίνησης και έχουμε μόνο μεμονωμένα περιστατικά που βεβαίως τα παρακολουθούμε εκ του σύνεγγης. Ε, το, το κλειδί για την εξέλιξη αυτή ήταν η εφαρμογή της διμερούς συμφωνίας Ιταλίας-Λιβύης στον τομέα ελέγχου συνόρων. Αυτό σαφώς επηρέασε τις εξελίξεις. Αυτό σημαίνει ότι τα βασικά μας μελήματα ε, επικεντρώνονται στα θαλάσσια σύνορα του χρόνου στο χώρο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Αυτό είναι το μεγάλο, αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν μιλάμε για παράνομη μετανάστευση, γιατί εκεί οι εξελίξεις ήταν κάπως θετικοί αλλά ε, όταν πρόκειται για ε, σοβαρότητα των ε, ροών αυτών είναι ενισχυτική η κατάσταση. Άλλος κοινός παρονομαστής, αν συγκρίνουμε Κανάρια, νησιά, Κεντρική Μεσόγειο και Ανατολική Μεσόγειο. Η Ανατολική Μεσόγειο στα σύνορα δηλαδή Ελλάδας-Τουρκίας, εκεί δεν έχουμε ε, διαρθρωτική, διαρθρωτική συνεργασία με την τρίτη χώρα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ε, θέμα και μια μεγάλη πρόκληση για τη Frontex που πρέπει να διαπραγματευτεί και να καταλήξει σε μια συνεργασία μεταξύ Frontex και Τουρκίας εις ό,τι αφορά τον έλεγχο των συνόρων. Δουλεύουμε πολύ σκληρά σε αυτό το τομέα επίσης. Τώρα, τα ανατολικά χερσαία σύνορα, πάλι η ανατολική οδός από την κεντρική Ασία, Ρωσία, Ουκρανία, Μολδαβία, Ουκρανία, μέχρι τις χώρες της κεντρικής ανατολικής Ευρώπης, κεντρικής Ευρώπης, ε, ήταν πολύ σημαντική οδός δεν το είπα, αλλά ίσως το είδατε στην προηγούμενη διαφάνεια, ότι οι τάσεις και τα, οι αριθμοί στα χερσαία σύνορα μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας και μεταξύ, στα χερσαία σύνορα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, εδώ οι αριθμοί είναι σχετικά υψηλοί. Όμως μπορείτε να δείτε πώς και πού ε, ασκούνται πιέσεις ε, στα χερσαία σύνορα ε, των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. Θέλω να αναφέρω και ορισμένα ε, θέματα σημαντικά στα χερσαία σύνορα και στα δυτικά ε, ε, στην Ανατολική Ευρώπη και στα Δυτικά Βαλκάνια που αφορούν τις ψευδείς αιτήσει ασύλου. Ένα κεντρικό θέμα είναι αυτό που το παρακολουθούμε και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε περισσότερο για να είμαστε βέβαιοι. Ποια είναι η ηθαγένεια των ε, προσφύγων όταν έχουμε αμφιβολίες σχετικά με την ορθότητα των στοιχείων που μας υποβάλλονται. Δηλαδή στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας ε, λιγότερο από το 10% των ε, μεταναστών έχουν στην πραγματικότητα την ηθαγένεια που δηλώνουν. Οπότε αυτό μας απασχολεί πάρα πολύ. Και θέλουμε να βρούμε τρόπους μέσα για να έχουμε μεγαλύτερη βεβαιότητα σχετικά με την προέλευση των ανθρώπων αυτών. Επανέρχομαι στη γενική ανασκόπηση των αποτελεσμάτων του 2009. Τώρα ε, έχουμε πολύ μεγαλύτερη επίγνωση των τεκτενομένων στα εξωτερικά σύνορα, που είναι οι προκλήσεις, γιατί συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν, τι κρύβεται από πίσω, πώς λειτουργούν ως επιτοπλίστων, πώς ε, δραστηριοποιούνται οι εγκληματικές οργανώσεις. Τώρα ξέρουμε πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι παλιά. Ένα πολύ σημαντικός δείκτης είναι ο αυξανόμενος αριθμός των εντοπιζομένων διακινητών. Αυτό είναι κάτι που ε, το κοιτάξαμε πολύ προσεκτικά, όχι μόνοι μας, αλλά μαζί με τις υπηρεσίες των κρατών μελών, δηλαδή συνοριακούς ελέγχους και την Europol για να εντοπίσουμε αυτούς που εκμεταλλεύονται τους παρανόμους, ε, τους παρανόμους μετανάστες. Ε, έχουμε δει ε, πώς λειτουργούν και έτσι μπορούμε με λιγότερες επενδύσεις να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, περισσότερες επιτυχίες. Θα επανέλθω σε αυτό. Ξέρουμε ότι ο έλεγχος των συνόρων δεν είναι από μόνος του ή μόνος του το κλειδί για την επιτυχία, αλλά βλέποντας τις επιτυχίες στα Κανάρια νησιά, στην Κεντρική Μεσόγειο, στα στενά του Γεβραλτάρ του συνοριακούς ελέγχους και τις ε, κοινέ επιχειρήσεις που συντονίσαμε, ε, βλέπουμε ότι έπαιξαν το ρόλο τους ε, για τις θετικές αυτές εξελίξεις. Αυτή είναι μια γενικότερη ανασκόπηση των αποτελεσμάτων του 2009 λοιπόν και τα πιο λεπτομερή στοιχεία θα υποβληθούν στην ετήσια έκθεση, έκθεση πεπραγμένων αργότερα. Οι προκλήσεις για το 2010 λοιπόν ε, θα είναι να παρακολουθήσουμε περισσότερο τις εξελίξεις και να έχουμε μεγαλύτερο επιχειρησιακό αντίκτυπο. Επίσης να αξιοποιήσουμε περισσότερο την τεχνική υποδομή των κρατών μελών. Και εδώ θα πω δύο λόγια αργότερα και όπως είπα υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες, αν υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες για την ηθαγένεια θα επικεντρωνόμεθα στο θέμα της, του εντοπισμού της πραγματικής ηθαγένειας. Αυτό είναι θέμα κλειδί. Γιατί αν δεν ξέρουμε από πού έρχονται οι άνθρωποι αυτοί, είναι πολύ δύσκολο να βρούμε και επαρκή μέσα για να λύμα. Όποια και αν είναι αυτά τα μέσα. Θέλουμε επίσης να συνεχίσουμε ε, στο τομέα της εναρμόνισης και θα πρέπει να είναι πιο διαλειτουργικές οι επιχειρήσεις μας, αυξάνοντας τη συνεργασία με τις, τρίτε τις τρίτες χώρες μεταξύ άλλων. Και αργότερα θα επανέλθω σε αυτό το θέμα της συνεργασίας με τρίτες χώρες. Ας προχωρήσουμε τώρα στην επιχειρησιακή ένταση. Αυτό με μεγάλη χαρά το δείχνω. Αυτή είναι η εξέλιξη των δραστηριοτήτων μας από το, που άρχισαν το 2006. Εμείς ε, πέρσι είμαστε λίγο μετριόφρονες όταν προσπαθήσαμε να προβλέψουμε την αύξηση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, αλλά εν τέλει μπορέσαμε να δούμε αύξηση 73% όταν πρόκειται δηλαδή για ημέρες επιχειρήσεων και από ε, μεταξύ 2009-2010 προγραμματίζομαι να ε, έχουμε αύξηση 24-25% της επιχειρησιακής έντασης. Οπότε έχουμε ακόμα ανεκμετάλλευτο δυναμικό και τις ικανότητες να ε, δραστηριοποιηθούμε περισσότερο σε αυτό το τομέα με την προϋπόθεση ότι και τα κράτη-μέλη θα ε, επιδείξουν ανάλογη βούληση. Η εκπαίδευση, κατάρτιση είναι πολύ σημαντικός τομέας, ε, το βάζω και αυτό για προβληματισμό και για λόγους σύγκρισης, να δείτε δηλαδή οι μέρες εκπαίδευσης, εκπαίδευσης που συντονίζονται από την Frontex και ποιες είναι οι προοπτικές για του χρόνου. Ήταν πολύ ε, σημαντική η εκπαίδευση και αυξήθηκε ε, δραστικά αυτό το δρόμο θέλουμε να ακολουθήσουμε, δηλαδή έτσι θα συνεχίσουμε και το 2010. Τώρα θα πω δύο λόγια για ε, τον τεχνικό εξοπλισμό, το crate το περίφημο, είναι, υπάρχει συνένωση. Δεν μιλάμε πια για toolboxes, εργαλειοθήκη. Αυτά εδώ είναι στοιχεία τωρινά των ε, εξοπλισμών και της υποδομής που έχουν τα κράτη-μέλη ιδιοκτησία τους και που μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε κοινέ επιχειρήσεις εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτουν τα κράτη-μέλη. Εδώ στηριζόμεθα στη βούληση των κρατών μελών, τα κράτη-μέλη δεν έχουν εντολή ούτε καμία υποχρέωση να αναπτύξουν τις δυνάμεις αυτές εάν δεν βλέπουν συντρέχει λόγος για κάτι τέτοιο. Ε, ένα κέριο μέλημα της Frontex σε αυτά τα πλαίσια αφορά το εξή. Περίπου 60% των επιχειρησιακών δαπανών της Frontex διοχετεύεται στην επιστροφή δαπανών των χωρών που φιλοξενούν την υποδομή αυτή, όχι των άλλων ευρωπαϊκών χωρών που συμμετέχουν στις ε, κοινέ επιχειρήσεις, οι μικτές επιχειρήσεις. Και ο στόχος μας το 2009 είναι να, ή το 2010 είναι να γίνουν πιο ευρωπαϊκές αυτές οι επιχειρήσεις, να συμμετέχουν και άλλα κράτη-μέλη στο σχετικά υψηλό επίπεδο δαπανών που επιστρέφονται στα κράτη-μέλη που φιλοξενούν αυτές τις υποδομές. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε υπόψη μας όταν ε, μιλάμε για την ε, διαχείριση του ενεργητικού, της υποδομής ε, στη διαχείριση της Frontex. Τώρα το Rabbit ε, ομάδες ταχείας επέμβασης στα σύνορα. Δεν υπάρχουν μεγάλες αλλαγές εδώ και δεν υπάρχουν διαφορές σε σχέση με το κανονισμό από το 2007. Κατεπίγουσες, έκτακτες ε, περιπτώσεις δεν είχαμε πολλές και γι' αυτό είχαμε κατάρτιση και ασκήσεις ε, ώστε το Rabbit να είναι ε, έτοιμο πόλεμο αν θέλετε και να μπορεί να αναπτυχθεί αν υπάρξει περιστατικό ανάγκη. Δύο ασκήσεις το χρόνο είχαμε προβλέψει, ναι, Ετησίω, το, από το 2007. Αυτό έγινε και το 2009, αλλά και το 2010 έτσι θα κάνουμε. Θα γίνουν δηλαδή τέτοιου είδους ασκήσεις, ούτως ώστε να δοκιμάσουμε την ετοιμότητα των κρατών μελών ε, να αναπτύσσουν ε, προσωπικό για αυτούς τους τομείς. Δύο λόγια τώρα για τις... Ε, επιχειρήσεις στα θαλάσσια σύνορα. Αυτή είναι η εικόνα για το 2010. Έχουμε μόνιμη υποδομή, έχουμε δίκτυο περιπολιών ευρωπαϊκών, ευρωπαϊκό δίκαιο, ε, δίκτυο συγγνώμη. Τα κράτη-μέλη συνδιοργανώνουν τις καθημερινές τους επιχειρήσεις και έχουμε εδώ κωδικούς ονόματα, δηλαδή κωδικών ε, που ανταποκρίνονται στις ε, φούσκες ή στα ε, βέλη αυτά. Ε, στα Κανάρια νησιά έχουμε. Ε, αυτά θα τα είναι κοινέ επιχειρήσεις που θα τις, προχωρήσω, θα τις προσπεράσω κάπως γρήγορα. Η Ήρα, Κανάρια νησιά, από τον Απρίλιο μέχρι τον Δεκέμβριο, όμως θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι τα προηγούμενα έτη η Ήρα, το πρόγραμμα Ήρα ε, παρατάθηκε μέχρι τον Απρίλιο του 2010. Τώρα, για την κεντρική Μεσόγειο και το χρόνο ως κοινή επιχείρηση είναι κωδικά, κωδικές ονομασίες, η Ήρα Κρόνος, αυτών των, κωδικές ονομασίες αυτών των επιχειρήσεων. Ε, από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο είναι ο χρόνος, γιατί εκεί είναι η ε, περίοδος εχμής ανάλογα με την ανάλυση και τα ιστορικά δεδομένα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι συμπεριλάβαμε στην ε, ε, ε, βοήθεια πριν από την επιστροφή στοιχεία που μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε μετά ολόκληρη τη διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολλοί εμπειρογνώμονες που θα ενημερώνουν, θα παίρνουν συνεντεύξεις από τους πρόσφυγες. Ο Ποσειδών, Ελλάδα-Τουρκία, θαλάσσια σύνορα. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό τρέχουσα περίοδο. Λαμβάνοντας υπόψη και τα, την παράταση ε, της λειτουργίας ε, πέραν του 2009, ε, θεωρούμε ότι θα συνεχιστεί αμύωτη διαδικασία αυτή το 2010. Καταμερισμός των πόρων, μην εκπλήσεστε και σοκάρεστε, θέλαμε μείωση περίπου κατά 10 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μια μείωση μείων 26% ε, για τις θαλάσσιες ε, ε, επιχειρήσεις. Μη φοβάστε όμως, μπορούμε παρόλα αυτά να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα για διάφορους λόγους. Μεταξύ άλλων μπορούμε τώρα να καταρτίζουμε ακριβέστερο προϋπολογισμό και με πιο αξιόπιστο τρόπο να κοστολογούμε αν θέλετε τις δαπάνες, οπότε πλέον οι υποχρεώσεις και οι πληρωμές αρχίζουν να ισορροπούν. Μπορούμε περισσότερο να προγραμματίζουμε τις ε, επιχειρήσεις αυτές με τις ε, την κατάρτιση, την επιστροφή, ούτως ώστε να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε με καλύτερο τρόπο από άποψη κόστους ωφέλους και επίσης τα μεταφερόμενα κονδύλια από έτος σε έτος, τα carry-overs, ήταν ε, ένα θέμα που μας απασχολούσε παλιά στις θαλάσσιες επιχειρήσεις. Εκεί επίσης έχουμε βελτίωση. Τώρα δηλαδή έχουμε καλύτερα αποτελέσματα με λιγότερα χρήματα. Αυτό είναι το σημαντικό. Χερσαίες επιχειρήσεις πάλι έχουμε μόνιμη δομή που είναι αυτά τα ε, ε γραφεία, ε, τα εστιακά, σε εστιακά σημεία τα οποία στελεχώνονται με μόνιμο προσωπικό λίγο πολύ και αυτά είναι τα κωδικά Jupiter, Neptune, Poseidon, δηλαδή ο Άρης, ο Κρόνος, ο Ποσειδόν Έχουμε ε, σαν εφεδρεία το Mars τον Άρη, JO Mars, Joint Operation. Αυτό μπορούμε να το αξιοποιήσουμε ε, αυξάνοντα ε, ε, τον αριθμό των εμπειρογνωμόνων ή των υποδομών που χρησιμοποιούνται αλλού, όπου κρίνουμε. Ε, Jupiter Poseidon, εδώ είναι τα, αυτά είναι τα βασικά, οι βασικές επιχειρήσεις, θα πρέπει να κλιμακώσουμε εδώ. Ένα αερίες επιχειρήσεις σχεδόν μόνιμες. Έχουμε τρεις διαφορετικές αντιλήψεις που έχουμε εδώ. Καταρχήν παρακολουθούμε τη ροή των επιβατών εδώ είναι τα προγράμματα Hammer και Hubble, επικεντρώνουμε σε επικεντρωνόμεθα σε κεντρικά αεροδρόμια ξένων χωρών για να παρακολουθήσω παρακολουθήσουμε τυχόν προβλήματα στις εναέριες ε, διαδρομές και έχουμε και εδώ το Meteor το οποίο είναι και αυτό μιας μορφής εφεδρεία που αποφασίζουμε πώς θα χρησιμοποιηθεί και στα αεροδρόμια έχουμε μόνιμη δομή επίσης και τα αισθιακά αυτά σημεία. Τώρα, ε, να δούμε και εδώ την κατανομή, στασιμότητα, στις χερσαίες, στασιμότητα και στις ενέργειες επιχειρήσεις. Και εις ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις επιστροφών, εδώ από άποψη δημοσιονομική θα έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση. Ένας λόγος είναι ότι έχουμε αυξημένες δραστηριότητες και το δεύτερο στοιχείο είναι η εσωτερική χρήση των διαφόρων δημοσιονομικών μέσων. Θέλουμε τώρα να χρηματοδοτήσουμε περισσότερο αυτές τις μικτές ή κοινέ ε, επιχειρήσεις επιστροφών από τον προϋπολογισμό μας. Θέλουμε επίσης να επεκτείνουμε στα κράτη-μέλη την ε, ε, ενίσχυση για τις επιστροφές, την υποστήριξη. Θα αναβλώνουμε αεροσκάφη από την Frontex για να τα χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη και αρχίζουμε με μικρότερα ε, αεροσκάφη όταν πρόκειται για τις ικανότητες και το έργο των σύνοριοφυλάκων και εδώ, αυτός είναι στόχος ε, κατάρτισης, να έχουμε καλύτερη κοινή κατανόηση θεμάτων ε, που έχουν να κάνουν και με τα θεμελιώδη δικαιώματα όταν πρόκειται για τέτοιου είδους επιχειρήσεις και θέλουμε μεγαλύτερη δραστηριοποίηση και σε επίπεδο κρατών μελών ή ε, κατανομή των των πόρων στις επιχειρήσεις επιστροφών βλέπουμε μία αύξηση σημαντική εδώ σε σχέση με πέρσι, δηλαδή με πέρσι το 2008. Ε, αυτό είναι μία από τις επιπτώσεις των αποφάσεων που ελάβαμε. Και θα προσπαθήσω να είμαι συνεπής. Δεν μιλάω για κατάρτιση και την ε, κατανομή των πόρων στην κατάρτιση και στις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης. Τα επίπεδα είναι ε, τα ίδια. το προσωπικό θα με το προσωπικό μας κατά 19%, πράγμα που σημαίνει ότι στο τέλος του 2010 Είμαστε περίπου κοντά στο, πιο κοντά στο 300. Ε, τα οικονομικά μας, δημοσιονομικά μας θα, είναι πολύ, θα βασίζονται σε αυστηρούς κανόνες. Ο προϋπολογισμός ε, για το 2010 είναι μειωμένο σε σχέση με πέρσι, αλλά το καλό είναι ότι τα δύο τρίτα μπορούμε να τα διοχετεύουμε των κονδυλίων για τις επιχειρήσεις και ένα τρίτο ε, καλύπτει διοικητικές δαπάνες. Αυτή είναι η εικόνα, να δείτε δηλαδή πώς μοιράζομαι, καταμερίζομαι τον προϋπολογισμό για τις διάφορες επιχειρήσεις. Ένα κεραίριο θέμα για του χρόνου είναι τα εξειδικευ... εξειδικευμένη κλάδη του Frontex για το, αυτό θα το κρίνει και το Διοικητικό Συμβούλιο. Έχει γίνει μια μελέτη σκοπιμότητας ήδη και έχουμε τώρα ένα σχέδιο σχετικά με το πώς θα γίνουν όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα λάβει τη σχετική απόφαση. Η δε ιδέα είναι να μπορούμε να έχουμε τέσσερα περιφερειακά γραφεία του οργανισμού Frontex τα επόμενα έτη, δηλαδή μέσα στην επόμενη τριετία. Θα ξεκινήσουμε προφανώς με μικρά έργα, πιλωτικά, βάσει και τις εμπειρίες που έχουμε και θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε στο μέλλον. Θα σταθούμε σε επιχειρησιακές δράσεις, πληροφόρηση και διαχείριση. Στόχος μας είναι να υπάρξει περιφερειακή κάλυψη. Η συνεργασία με τις τρίτες χώρες και αυτήν την τελευταία διαφάνεια ε, πολύ σημαντική, αλλά παρακαλώ την υπομονή σας. Έχουμε 12 συμφωνίες εργασίες που λειτουργούν με τρίτες χώρες, όλες γειτονικές, στα ανατολικά σύνορα, ε, Ρωσία, Λευκορωσία, Μολδαβία, Ουκρανία, που παίζουν όλες βασικό ρόλο στις επιχειρησιακές δραστηριότητες της ε, ε, Frontex. Το ίδιο συμβαίνει και με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων με τις οποίες έχουμε μια συμφωνία που λειτουργεί. Ε, προσπαθούμε να πετύχουμε τη συμφωνία με την Τουρκία. Αυτό είναι προτεραιότητα στις συνεργασίες με τρίτες χώρες και βεβαίως συνεχώς προσπαθούμε να έχουμε μια θετική εξέλιξη στις διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο, την Τινησία, τη Λιβύα και την Αίγυπτο. Και εδώ τελειώνω πραγματικά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Κύριε Λάτινεν, καλύψατε και το σημείο 5 της ημερής διάταξης, έτσι. Ερωτήσεις. Έξι άτομα έχουν ζητήσει το λόγο, επτά, οκτώ, πολύ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, γιατί πρέπει να συζητήσουμε και το σημείο 6. Και όλα αυτά πρέπει να λήξουν σε μισή ώρα περίπου. Δεν ξέρω γιατί. Ε, πέντε είναι η ψηφοφορία. Η γραμματεία γιατί μας λέτε ότι... Α, έχουμε ναι και τις ε, θεωρήσεις ε, μακράς διάρκειας. Μισή ώρα συνολικά. Θα ήθελα λοιπόν να περιοριστείτε σε ερώτηση ενός λεπτού. Να μην κάνετε δηλώσεις για να υπάρξει μια χρόνος για συζήτηση. Η κυρία Μποσελίνο. κυρία αλλά δεν σας βλέπω. Πέρσι ήσασταν ο κύριος Λαμπρινίδης. Ευχαριστώ κύριε Λάτιν που ήρθατε. Δύο πολύ σύντομες ερωτήσεις. Πρώτον, αύξηση δραστηριοτήτων για το 2010 οι περισσότερες δραστηριότητε αφορούν πιλωτικά έργα, όχι επιχειρήσεις. Η ερώτησή μου είναι τι είναι αυτά τα πιλωτικά έργα που προγραμματίζεται για το 10. Δεν τα σχολιάσατε παρκώς. Δεύτερον, διαπραγματεύσεις με την Τουρκία. Μπορείτε να μας εξηγήσετε κάπως καλύτερα πώς προχωρούν. Όλοι γνωρίζουμε ότι πολλά ελικόπτερα της Frontex και άλλες δραστηριότητες στην περιοχή δέχθηκαν μηνύματα από τουρκικές αρχές που σχετίζονται με το ότι θεωρήθηκε ότι, ότι παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Τουρκίας. Αυτό μου δημιουργεί ανησυχία το ότι ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν οι διαπραγματεύσεις αυτές όχι για το στόχο τους, δηλαδή να βοηθήσουν την Ευρώπη να προσπίσει καλύτερα τα σύνορά της, αλλά από την παράνομη μετανάστευση, αλλά για να θετεθούν ε, ζητήματα για την κυριαρχία της Ελλάδος, κάτι που έχει γίνει από πλευρά του Τουρκία στο παρελθόν. Μπορείτε να μας πείτε λίγα περισσότερα πράγματα γι' αυτό, πώς προχωρούν οι διαπραγματεύσεις, έχετε αντιμετωπίσει τέτοια ζητήματα, τι συνεργασία έχετε με την ελληνική κυβέρνηση σήμερα για να εξασφαλίσετε την βέλτιστη δυνατή συνεργασία και συντονισμό στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Βλέπω ένα ρολόι, δεν ξέρω αν το βλέπετε όλοι. Δεν μπορείτε. Θα σας εξετάζω αναομάδες 5. Η, κύριε Λάτφορντ κατόπιν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λάτιναν. Οι δραστηριότητε Frontex σας έδωσαν βάση για να δώσετε στην Επιτροπή σε και στο Συμβούλιο απαντήσεις σε τομέα πολιτικής. Είδα το κείμενό σας για τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στην μετανάστευση των ελίτ. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Εκεί αναφέρεται ότι οι περιορισμοί στην μετανάστευση στην Ευρώπη που ξεκίνησαν από το 1973 και συνεχίστηκαν από το 80, στη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90 θεωρούνται από πολλούς ως η πηγή των ε, ε, καταχρηστικών ετοιμάτων ασύλου. Και ότι μια πολιτική και υποστηρίζεται μια πολιτική νόμιμης και μόνιμης μετανάστευσης. Είπατε επίσης ότι οι πιέσεις στα ελληνοτουρκικά σύνορα είχαν ήταν ε, συνέπεια της συμφωνίας μεταξύ Ιταλίας Λιβύης. Παρακολουθείτε τι γίνεται στη Λιβύη. Αναφέρεται ότι η στόχη της Frontex κλείνεται, κλείνεται λέει πρόεδρος. Ναι, θέλω να πω ότι εξασφαλίζεται ότι αυτοί που επιστρέφεται την χάνουν δίκαιης αντιμετώπισης σε ό,τι αφορά τα δικαιώματά τους. Δεν έχουμε χρόνο, λέει η πρόεδρος, ο κύριο Μωράς και μετά η κυρία Κέλλερ. Θα είμαι σύντομος. Ήθελα να θέσω τα βασικά ερωτήματα που θα έρθουν στο επόμενο θέμα, ε, τον κώδικα με σύνορων Σέγγεν, διότι οι αποβιβάσεις, για παράδειγμα, είναι θεμελιώδη. Κάποια από αυτά τα υπέρ ανέφερε η κυρία Λάτφορντ. Θα Δεν θα μιλήσω γι' αυτά. Σε ό,τι αφορά τη Frontex, είχαμε κάποιες συζητήσεις με την Επιτροπή για τα επιχειρησιακά στοιχεία της Frontex. Έχετε κάποια πάγια στοιχεία ή εξαρτάστε μόνο από τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι θεμελιώδη στοιχείο. Είπατε επίση ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί. Αλλά αυτό εξαρτάται από την καλή πρόεδρεση του καθενός. Πώς είναι η κατάσταση. Υπάρχουν κράτη που είναι πιο καλά, πιο επιμελή από άλλα σε ό,τι αφορά την παροχή στοιχείων, στοιχείων ενεργητικού. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, το χρόνο τον βλέπετε στο μηχάνημα, στο μηχάνημα ψηφοφορίας. Η κυρία Κέλλερ, η κυρία Κλάς και μετά ο κύριος Λάιτεν θα απαντήσει. Ευχαριστώ θα επεκταθώ σε αυτά που είπε η κυρία Λάτφορντ. Τι συμβαίνει με αυτού που επιστρέφεται, ξέρετε, σε όλε τι χώρε, όχι μόνο τη Λιβύη. Μετά αναφέρεται ότι ένα από του στόχου τη Frontex είναι να υπάρξει κοινή κατανόηση για την ανάπτυξη των, των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων Frontex. Το πετυγχάνεται αυτό. Επίση, υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες υπήρξε επαναπροώθηση από πλευράς ε, ε, εργαζομένων στη Frontex. Τελευταία ερώτηση, προπολογισμό. Ο προπολογισμό δεν ανταποκρίνεται στην ιδέα που δώσετε ότι 50% των ατόμων παίρνουν από τα χερσαία σύνορα. Τα περισσότερα κονδύλια σας τα δαπανάτε στη θάλασσα, στα θαλάσσια σύνορα. Πώς το εξηγείτε αυτό. Είναι ακριβότερο να γίνεται διάσωση στη θάλασσα ή γιατί υπάρχει αυτή η αναντιστοιχία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κλάς και μετά ο κύριος Λάιτενεν θα απαντήσει. Δύο λεπτά θα έχει ο κύριος Λάιτενεν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Λάιτινεν, έχω μία ερώτηση, μία ιδιόμορφη ερώτηση αν θέλετε, σε μία χώρα που πολύ κομψά ορίσατε ως τρίτη χώρα. Μα εδώ δεν πρόκειται όμως για τρίτη χώρα, για υποψήφια χώρα πρόκειται, για την Τουρκία μιλάμε. Εδώ και πολλά χρόνια το Frontex ε, ε, επισημαίνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στη συνεργασία μας με την Τουρκία, που είναι όχι απλά και μόνο χώρα προέλευσης, αλλά είναι χώρα διαμετακόμισης μεταναστών. Πρόκειται λοιπόν για μια χώρα υποψήφιο πρέπει να την αναγκάσουμε ούτω να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Ρωτώ λοιπόν, τι εξελίξεις προβλέπετε, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα για την εξέβρεση συμφωνίας. Ευχαριστώ. Γκρινιάζετε συνάδελφοι, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι εκεί που, από εκεί που προέρχομαι εγώ έχουμε κάθε ώρα μόνο 60 λεπτά. Δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Δεν, δεν έχουμε ώρα παραπάνω από 60. Έχουμε μισή ώρα, τελείωσε. Ίσως να μας βοηθήσει ο κύριος Κοέλιο, κύριε Μπουσούτιλ. Θα έρθει πάντως. Θα έχουμε, εάν φάμε μισή ώρα εδώ, θα έχουμε 20 λεπτά για τη συζήτηση του άλλου του σημείου 6 πριν την πληροφορία στις 5. Το μόνο που μπορώ να ζητήσω είναι να είναι σύντομος ο κύριος Λάτινεν. Μιλήσετε πάρα πολύ. Ε, τόσα κάνουμε, τόσα μπορούμε. Θα γκρινιάζουν όλοι. Επί της διαδικασίας ο κύριος Μπουσούτιλ. Διαμαρτύρομαι πρόεδρε. Δεν πρέπει να γίνονται έτσι τα πράγματα. Πρόκειται για μια ευκαιρία, σπάνια ευκαιρία. Ο κ. Λάτινεν δεν έχει έρθει εδώ και καιρό. Πρέπει να έχουμε μία σειρά λεπτομεριακών απαντήσεων στις ερωτήσεις που θέτουμε. Εξού, γι' αυτό υπάρχει και η συνάντηση. Είχαμε πει ότι οι συνεδρίες θα κρατούσε μέχρι τις 5. Γιατί να χάσουμε 15 λεπτά από το χρόνο μας τώρα, κύριε Μπουσουτήλ. Ήσασταν εδώ όταν εγκρίναμε την ημερήσια διάταξη. Δεν την έφτιαξα εγώ την ημερήσια διάταξη. Έφυγαν κάποια σημεία και έχουμε αυτό το χρόνο. Ε, έτσι είναι η ζωή. Δεν το επέλεξα εγώ αυτό. Παρακαλώ κύριε Λάιτινεν να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι εξαιρετικά σύντομος. Να απαντήσω από κοινού σε κάποιες ερωτήσεις. Πρώτον, προτεραιότητες. Η συμφωνία με την Τουρκία η συνεργασία με την Τουρκία. Δεν έχουμε καμία ψευδέστηση ότι η συνεργασία μεταξύ κρατών μελών της Ένωσης και της ε, τρίτης χώρας αυτής θα λύσει τα πολιτικά ζητήματα. Δεν αντιμετωπίζουμε, δεν εξετάζουμε πολιτικά ζητήματα, μιλούμε μόνο για επιχειρησιακά ζητήματα. Φερρυπίν, πώς θα γίνει ανταλλαγή πληροφοριών και πώς θα συγκρίνουμε την ανάλυση κινδύνου, πώς θα συνεργαστούμε στον τομέα της κατάρτισης, της έρευνας και ανάπτυξης και το πώς οι συνάδελφοι ε, από τις δύο πλευρές των συνόρων θα μετέχουν στις κοινέ ε, ε, δραστηριότητες. Αυτό είναι η βάση της ε, συμφωνίας ε, συνεργασίας μεταξύ της Frontex και όλων των τρίτων χωρών και αυτό συμβαίνει και με την Τουρκία. Οι διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο βρίσκονται σε τελική φάση. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν πάρα πολύ σύντομα. Επίσης, γνωρίζουμε το ενδιαφέρον και τις ανησυχίες των διαφόρων κρατών μελών και των ευρωπαϊκών οργάνων και παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά τις σχετικές εξέλιξεις. Πιλωτικά σχέδια. Κάποιοι, στην πραγματικότητα πρόκειται συνήθως για δοκιμές νέων μοντέλων. Ευρωπαϊκές περιπολίες για παράδειγμα ήταν ένα μοντέλο. Ε, η κοινή, η κοινή επιχείρηση Hubble και αυτό ήταν πιλωτικό σχέδιο όταν το δοκιμάζαμε πριν γίνει επιχειρησιακή δράση. η μετακίνηση από Ιταλία στη Λιβύη. Παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς τις συνέπειες της ε, τις συνέπειες ε, της μετακίνησης των, της απομάκρυνσης προς τα εκεί. Όταν προχωρούμε στην εφαρμογή της διμερούς, ε, διμερών συμφωνιών μεταξύ κράτους μέλους της Ένωσης και τρίτης χώρας, η Frontex δεν μπορεί να προχωρήσει σε οποιαδήποτε έρευνα για το τι γίνεται δεν είμαστε ερευνητικό οργανισμό ούτε έχουμε τι αρμοδιότητε. Ό,τι μαθαίνουμε, όταν μαθαίνουμε ότι κάτι συνέβη, προσπαθούμε να δούμε τι έγινε, προσπαθούμε να βρούμε περισσότερες πληροφορίες και αν βρούμε ότι κάτι υπάρχει, το αναφέρουμε στο αρμόδιο ευρωπαϊκό όργανο που ασχολείται με την επιβολή, με, με την εφαρμογή του νόμου. Ε, τώρα, κατανομή των πόρων. Προφανώς είναι ακριβότερες οι ε, δραστηριότητε στη θάλασσα, χρησιμοποιούμε βενζίνη, πετρέλαιο δηλαδή για τις μηχανές, ε, σκάφη. Ε, το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο, 6.000 ευρώ την ώρα, από, ενώ αυτό δεν συμβαίνει στα χερσαία σύνορα. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η αναντιστοιχία. συμμετοχή κρατών μελών στις κοινέ επιχειρήσεις. Έχουμε θετικές εξελίξεις στην συμμετοχή τους. Μπορέσαμε να αυξήσουμε τις επιχειρησιακές δραστηριότητε. Θέλω να τονίσω ωστόσο ξανά ότι 60% των, του προπολογισμού των επιχειρήσεων Frontex καλύπτουν σύγχρηματοδοτούν δραστηριότητε της χώρας υποδοχής, της, της φιλοξενούσας χώρας, συγγνώμη. Και αυτό είναι κάτι που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και που πρέπει να αντικατοπτρίζεται όταν ξεκινήσει η συζήτηση για την αγορά ε, περιουσιακών στοιχείων της Frontex. Επειδή να κάλυψε όλα τα βασικά ζητήματα, σύντομα. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Άλλοι οκτώ συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ να είστε σύντομοι. Η κυρία Χένη και η κυρία Αλβάρο. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη. Τουρκία. Και εμεί το ίδιο μήνυμα είχαμε, είχαμε πάρει το ίδιο μήνυμα και πέρσι. Ότι θα ολοκληρωθούν οι συμφωνίε συνεργασία με την Τουρκία. Τι εμποδίζει την Τουρκία από την υπογραφή. Είπατε το ίδιο πράγμα και πέρσι. Το ίδιο λέτε και τώρα για τα περιουσιακά στοιχεία της Frontex και την αντιστοιχεία των δαπανών. Συμφωνείτε να υπάρξει ένας μηχανισμός δεσμευτικός προς τα κατημέλη για να μετέχουν στην, στις δαπάνες και στην περιουσία του Frontex, στο ενεργητικό δηλαδή. Και πιστεύετε ότι μια συμφωνία που θα περιέχει τις βασικές γραμμές του, του δικαίου της θαλάσσια θα βοηθούσε, η κύρια Αλβάρο. Εγώ να ρωτήσω το εξή στον κύριο Λάιτενεν. Μίλησε για αλληλεγγύη και ανθρωπισμό στο Frontex και μετά μας μίλησε για τον χρόνο. Λέγοντας ότι στην στα πλαίσια του χρόνου έχει παρισφρήσει συμφωνία μεταξύ Ιταλίας και Λιβύη. Τι γίνεται όμως, πώς μπορούμε εμείς να μιλάμε για ανθρωπισμό και, και ανεκτικότητα όταν έχουμε την, την, την επαναπρόθεση όλων αυτών των προσφύγων στην Λιβύη και πώς αντιμετωπίζετε αυτή τη διμερή συμφωνία όταν η Ευρώπη ετοιμάζεται να διαπραγματευτεί με τη Λιβύη. Ξέρετε κάτι σχετικά. Ο κύριος Μπουσούτιλ για το κράτερο. Φέτος θα γίνει αναθεώρηση της εντολής του οργανισμού. Εσείς θα συμβουλεύσετε να μετατραπεί ο θελοντικός χαρακτήρας συμμετοχής στο κρέιτερ σε δεσμευτική υποχρέωση για τα κρατημέλη, όχι. Δεύτερον, μιλήστε για το Rabbit. Ε, υπάρχει νομοθεσία, αλλά που δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ. Κατά την άποψή σας, αυτό είναι μια μάταιη πρωτοβουλία ή μπορεί ή πώς μπορεί να γίνει ε, επιτυχής. Ευχαριστώ πρόεδρε δύο ερωτήσεις για την σελίδα 2 της διαφάνειάς σας. Αναφέρει ότι το 2009 167.700 άτομα, αύξηση 22%. Αυτή είναι αυτή που είδε η Frontex όμως. Αυτή που δεν είδε η Frontex, ωραίο είναι να βλέπεις. Αλλά τι έχετε να μας πείτε για αυτούς που δεν βρήκατε. Δεύτερη ερώτηση. Λέγεται παράνομη διέλευση των συνόρων και άρνηση εισόδου. Το δεύτερο είναι κάτι το επίσημο. Ενώ η παράνομη διέλευση συνόρων είναι παράνομη εξορισμού. Ποια είναι η διάκριση μεταξύ των δύο κατηγοριών αυτών. Πόσοι υπάγονται στην άρνηση εισόδου και πόσοι είναι παράνομοι διέλευση συνόρων. Η κυρία Φλότρο και μετά ο κύριο Λάιτινεν. Αν κατάλαβα καλά, εσείς είπατε ότι κατά τις εκτιμήσεις σας ένα 10% άλλο δαπών ή να το πω καλύτερα είναι μόνο το 10% αυτών των παρανόμων στην Τουρκία που δηλώνουν την πραγματική τους υπηκότητα. Αυτό είπατε, το επιβεβαιώνετε. Και μετά είχατε ιδιαίτερε υπεκφυγέ, χρησιμοποίησατε ιδιαίτερε υπεκφυγέ όταν μιλούσαμε για διεθνεί προδιαγραφέ και διεθνεί συμφωνίε, ε, για τη συμφωνία τη Γενέβη, ε, για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Μπορείτε να μας πείτε πώς το αντιλαμβάνεστε εσείς ο ίδιος αυτό το θέμα των υποχρεώσεων που έχουμε στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου και το πώς το αντιμετωπίζει ο οργανισμός που εσείς διευθύνετε. Και επίσης ε, τι προβλέπετε στο πρόγραμμα του 2010 και στα οικονομικά σας αιτήματα ε, ως χρηματοδότηση για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τις απαιτήσει του διεθνούς δικαίου, ο κύριος Λάιτινεν. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Πάλι θα αρχίσω με την Τουρκία και τις ε, ρυθμίσεις που έχουμε προβλέψει. Χρειάζεται να συνεργαστούν και τα δύο μέρη εδώ. Δεν μπορεί να υπαγορεύσει ο ένας και να συμφωνήσει ο άλλος θα πρέπει να δούμε τι συμφωνία θα είναι αυτή και πώς θα συνεργαστούμε μέχρι εκεί. Έχουν προχωρήσει οι τεχνικής φύσεως συζητήσεις και φαίνεται ότι υπάρχει μια κοινή κατανόηση για το εύρος αυτό της συνεργασίας που είναι πολύ επιχειρησιακή, περιλαμβάνει δε αυτά που σας είπα, κατάρτιση, ανταλλαγή πληροφοριών, κάποιοι τομείς έρευνας και ανάπτυξης και πώς θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε όταν αρχίσουν να τρέχουν οι κοινέ επιχειρήσεις. Επιχειρησιακής φύσεως πράγματα. Δεν ε, πάμε να ε, αναμειχθούμε στα ανοιχτά ζητήματα που υπάρχουν σε αυτή την περιοχή να τα λύσουμε. Είμαστε πολύ πρακτικοί στην προσέγγιση μας. Τώρα, για τα στοιχεία του ενεργητικού μας, του ενεργητικού που υπάρχουν, ε, τι δεσμευτεί τι δέσμευση υπάρχει να έχουμε δικούς μας εξοπλισμούς. Δεν νομίζω ότι είναι σόφρον εξέλιξη να κάνουμε δραστικές κινήσεις ε, σχετικά με το πόσο δεσμευτική δηλαδή θα είναι η κοινή συμμετοχή των κρατών μελών στις επιχειρήσεις. Εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε αυτό που κάναμε και μέχρι τώρα, δηλαδή να ε, Έχουμε αυτή τη θετική ενθάρρυνση να δραστηριοποιηθούν σιγά σιγά, να έχουν χρόνο να δουν πώς αντιμετωπίζουμε τις ευρωπαϊκές προκλήσεις. Δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το μαστίγιο αντί για το καρότο. Όμως, παράλληλα θέλουμε και μια μεγαλύτερη ανεξαρτησία ώστε να μπορούμε να έχουμε την ε, ικανότητα αντίδρασης ε, και αυτό έχει σχέση με την ύπαρξη κάποιων στοιχείων του ενεργητικού δικά μας, της Frontex. Ε, μια υποδομή που θα μπορούμε να κινητοποιούμε αν συμβεί κάτι, αν κρίνουμε ότι κάποιοι εξοπλισμοί θα πρέπει να ε, κινητοποιηθούν, να χρησιμοποιηθούν σε κάποιες σημαντικές επιχειρήσεις. Θέλω λοιπόν μεγαλύτερη ενθάρρυνση των κρατών μελών για να συμμετέχουν περισσότερο στις κοινέ επιχειρήσεις και να μπορεί να δικαιούται δηλαδή, να νομιμοποιείται η Frontex, να έχει δικούς της εξοπλισμούς ως ένα βαθμό, ούτω ώστε να ε, εξασφαλίζεται αυτή η επιχειρησιακή ικανότητα. Τώρα για, για το Rabbit. Αυτό σκοπό είχε να είναι ένα μέσον ε, κατεπήγοντος έκτακτης ανάγκης. Γιατί? γιατί είναι δεσμευτική συμμετοχή εδώ στα, για τα κράτη-μέλη, οπότε το κατόφλιο για την ανάπτυξη, χρησιμοποίηση αυτών των εμπειρογνωμόνων ειδικών είναι υψηλό. Ε, έκτακτες ανάγκες, κατεπήγοντα κλπ. Μέχρι τώρα αυτές τις ασκήσεις τις είχαμε δύο φορές το χρόνο, πολύ καλές. Ε, συμμετείχαν περίπου 700 εμπειρογνώμονες σε αυτό το πουλ δυνάμεων και βέβαια υπάρχει λόγος γι' αυτό. Ξέρουμε έτσι πώς, θα, πώς λειτουργεί το σύστημα, αν χρειαστεί να κινητοποιηθεί. Και επίσης, σχεδόν όλοι αυτοί οι 700 εμπειρογνώμονες στο πουλ του Rabbit είναι μέλη και άλλου pool που είναι εθελοντικό, που είναι το FJST, που είναι το Frontex, το Κοινό Σύστημα Υποστήριξης. Και αυτοί είναι που μετέχουν και στις ε, τακτικές, στις κανονικές επιχειρήσεις, ε, περιοδικά και συστηματικά σε όλο το χρόνο. Τα μέλη Rabbit πάντοτε συμμετέχουν στις συνήθεις επιχειρήσεις της Frontex. Όταν πρόκειται τώρα για τις ασκήσεις και κατάρτιση Rabbit, θέλουμε να δοκιμάσουμε περισσότερο τις διαδικασίες και την δυνατότητα ταχείας ανάπτυξης αυτών των δυνάμεων, αν χρειαστεί, των δυνάμεων των εμπειρογνωμόνων. Δεν είναι δηλαδή ε, εναλλακτικά είναι τα συστήματα Rabbit και FJSC ε, είναι αλληλοσυμπληρωνόμενα. Ο κ. Μπραντεκα με έκανε μια πολύ εύστοχη ερώτηση σχετικά με το τι δεν ε, είδαμε. Μακάρι να μπορούσα να σας απαντήσω, γιατί αυτό είναι το Άγιο Δισκοπότηρο των δυνάμεων ε, καταστολής ε, σχετικά με το κρυφό έγκλημα. Τώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχουμε ακόμα καν ε, ούτε αξιόπιστες εκτιμήσεις σχετικά με το ποσοστό του κρυφού εγκλήματος. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό το θέμα, προσπαθώντας να επικεντρωθούμε περισσότερο στην αξιολόγηση των ευάλωτων σημείων των κρατών μελών, να βρούμε ένα δίκτυο, αν θέλετε, που θα μας επιτρέψει να με την αξιοπιστία των συστημάτων των κρατών μελών και των δικών μας κοινών επιχειρήσεων. Αλλά οπωσδήποτε αυτό θα πάρει δέκα χρόνια. Είναι ένα θεμελιώδες ερώτημα. Δηλαδή να μπορούμε να δούμε αυτό που είναι κρυφό, που δεν φαίνεται. Αυτά προς το παρόν ως απάντηση από την πλευρά μου. Α, ξέχασα κάτι Πρόεδρε, ήταν και η δικιά μου ερώτηση και δεν απαντήθηκε. Απαντήστε και σε αυτά σύντομα παρακαλώ. Ναι, για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Πολύ συχνά ε, πρέπει να δούμε αυτά τα ζητήματα, δηλαδή πώς θα πρέπει να αντιδρούμε σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ισχυρισμό ότι παραβιάστηκαν τα, ανθρώπινα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και πρέπει να είμαστε πολύ ειλικρινής σε αυτό το θέμα. Ο έλεγχος συνόρων πάντοτε ε, δημιουργεί τέτοια προβλήματα. Ε, υπάρχουν καταγγελίες. Θέλουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση μέσα από την ε, κατάρτιση, εντάσσοντας κάποια θέματα στα επιχειρησιακά μας προγράμματα, αλλά δεν μπορεί κανείς να πει ότι όλα τα προβλήματα μπορούν να λυθούν από αυτούς που ε, ασκούν τον έλεγχο των ε, συνόρων. Δεν ε, μπορούμε πολλές φορές να κάνουμε τις σωστές ανακρίσεις και έρευνες, θα κάνουν τα κράτη-μέλη. Έχουμε ένα σύστημα υποβολής εκθέσεων και αναφορών όταν... Ε, Επιχειρήσει είναι κοινέ και αν υπάρχει κάποια καταγγελία ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο, η ευρωπαϊκή νομοθεσία ή κάποια άλλη νομοθεσία έχουν παραβιαστεί και παραπέμπουμε τα θέματα αυτά στον αρμόδιο φορέα και πολλές φορές έχουμε απευθυνθεί, έχουμε παραπέμψει τα θέματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, είμαστε πολύ σοβαροί στην αντιμετώπιση αυτών των ε, θεμάτων, αλλά βεβαίως θα πρέπει να γίνει κατανοητός και ο δικός μας ρόλος εδώ. Και το ίδιο ισχύει και για τη συνεργασία μεταξύ ενός κράτους μέλους και μιας τρίτης χώρας, ε, Λιβύης και Ιταλίας ε, εν προκειμένου. Δεν μπορεί η Frontex να παίξει το ρόλο του κριτή και να πει ποιο το σωστό και ποιο το λάθος. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μας. Ιδιαίτερα ε, εφόσον δεν είμαστε εμείς εταίρος ή παίκτη, αν θέλετε, σε αυτές τις ε, καταστάσεις. Γενικά όμως, όταν πρόκειται για πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε μακροπρόθεσμη προοπτική, εκεί στοχεύουν η κατάρτισή μας και τα αναλυτικά προγράμματα κατάρτισης επικεντρώνονται σε αυτά τα θέματα και θέλουμε βεβαίως να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τα πράγματα μακροπρόθεσμα, μέσα από την κατάρτιση πάντα, ούτως ώστε να τα γνωρίζουν τα θέματα και να αντιδρούν οι συνοριοφύλακες ανάλογα. Ευχαριστώ. Και άλλοι τρει ομιλητές θέλουν να μιλήσουν. Εγώ θα πρέπει να φύγω. Βλέπω και ο κύριο είναι... Εγώ θα φύγω και θα δώσω αυτή βέβαια στον κύριο Γιακουλίνο. Έχω να πάω σε μια άλλη συνάντηση όπως σας είπα που ξεκίνησε. Ευχαριστώ τον κύριο Λάιτνεν ε, προς το παρόν. Ο κύριος Σταβάρες έχει διαδικαστικό. Μήπως θα έπρεπε να έχουμε τον κατάλογο των μιλητών στο ξεκίνημα. Εγώ ήμουν ο δεύτερος τρίτος που σήκωσε το χέρι του. Θέλω να ξέρω λοιπόν, γραφτήκαμε, όχι τώρα, εν γέννη. Εγώ σας βλέπω στο ξεκίνημα συνήθως. Ε, δεν μπορώ να πω ότι ε, είναι δυνατό, πιθανόν να σας ε, ε να μην σας είδα. Κάνω ό,τι μπορώ. Θα μας βοηθούσε και εμένα και εσάς αυτό πάντως πρόεδρε, λέει ο κύριος Σταβάρης. Αντικαταστήσω την συνάδελφο. Συνεχίζουμε τις δραστηριότητε και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι είχαν ζητήσει να λάβουν το λόγο. Ο κύριος Έντσου.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 υπήρχαν πόροι που δόθηκαν σε τρίτες χώρες και θα ήταν μια καλή ιδέα να υπάρχουν κοινέ έρευνε ή όχι. Και εγώ έκανα μια ερώτηση. Ε, σύντομη θα είναι. Η εξή. Μυρίσετε για τέσσερα βασικά στοιχεία, τέσσερις πυλώνες που διαπούν την δραστηριότητά σας. Μεταξύ αυτών η συμφωνία με τα κράτη-μέλη. Μετά είπατε ότι αυτό δεν λειτουργεί πάντα και είπατε ότι μερικές φορές τα ίδια εργαλεία που τίθεται στη διάθεση της Frontex χρησιμοποιούνται και από τις ε, χώρες μέλη. Ρωτώ, με, την πρόσφατη, με το πρόσφατο κείμενο της Στοκχόλμης ενισχύθηκαν οι αρμοδιότητες της Frontex. Βελτίωσε η πρωτοβουλία της Στοκχόλμης στην συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Πώς μπορείτε να λειτουργήσετε ως κινητήριος δύναμη χωρίς την, με, την ε, συμμετοχή των κρατομελών. Κύριε Σταβάρες. Καλό είναι να γκρινιάζει κανείς. Μας δώσατε, κύριε Λάτινερ, τα κονδύλια για τις θαλάσσιες επιχειρήσεις και είπατε ε, μην ανησυχείτε από την μείωση γιατί μπορεί να κάνουμε περισσότερα πράγματα με λιγότερα λεφτά. Εγώ μπορώ να σας πω πώς να τα χρησιμοποιήσετε. Δεν μιλάμε για μεταφορά υλικού, ε, άειλων προϊόντων, αλλά για ανθρώπους. Οι άνθρωποι αυτοί φεύγουν από περιοχές και από χώρες που ε, αντιμετωπίζουν ε, κρίση, που διώκονται. Ενδέχεται να είναι τούντες άσυλοι οι πραγματικοί πρόσφυγες. Θα ήθελα να ξέρω πώς εξετάζεται αν αυτοί οι άνθρωποι είναι ή όχι πρόσφυγες. Τι κάνετε, κάνετε συνεντεύξεις Μήπως οι πόροι που έχετε θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να ε, ελεγχθεί η πραγματική υπηκότητά τους και να καταπολεμηθούν οι καταχρηστικές ή ψευδείς δηλώσεις ε, για να καταλάβουμε και αν είναι οι άνθρωποι αυτοί πρόσφυγες ή όχι. Μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι δεν επιστρέφεται ποτέ κάποιος που κινδυνεύει να διωχθεί σε μια χώρα όπου μπορεί να υποστεί τον κίνδυνο αυτό. Μήπως η Frontex θα έπρεπε να ανοίξει τις αποστολές της και στην ύπατη αρμοστία του για τους πρόσφυγες. Και επίσης, αυτό είναι μια ευθεία ερώτηση. Πότε θα ανοίξετε τις δραστηριότητε, θα επιτρέψετε δηλαδή να μετάσχουν στις δραστηριότητε και εκπρόσωποι της ύπατης αρμοστίας. Κύριος Κοντσέτα, παρακαλώ. μιλήσατε στην ανάλυση σας στο γεγονός, αναφέρατε στο γεγονός ότι η Μεσόγειος, η περιοχή γύριος μεταξύ Ιταλίας, Μάλτας, Λιβύης, ε, είδε μία μείωση δραστηριοτήτων της Frontex που είναι άσχετες με την μείωση των θαλάσσιων εν γέννη δραστηριοτήτων. Άρα τι σημαίνει ότι εκεί δεν παρεμβαίνεται συγκεκριμένα. Η δική μου εικόνα είναι ε, ότι ουδέποτε υπήρξε παρέμβαση της Frontex. Δηλαδή ε, το θέμα των μεταναστευτικών ροών στην περιοχή αυτή ε, στην ουσία εκχωρήθηκε στις δύο χώρες, την Ιταλία και τη Μάλτα. Και ότι αυτό συνεχίζει να είναι έτσι από κάθε οπτική γωνία και θετικά και αρνητικά. Αυτό έχει συνέπειες και για τις διμερείς συμφωνίες που συνάπτουν ε, τα κράτη-μέλη με τρίτες χώρες. Εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Υπάρχει κοινό μέτωπο στα θέματα του ελέγχου των μεταναστευτικών ροών. Η υπάρχουν κοινέ πηγές που να ελέγχουν τις να, να, να παριθμούν τις ροές και τα λοιπά. Και ξέρουμε τα σχετικά με τις διαδρομές μπορεί κάποιος να μπει στην Ελλάδα και να καταλήξει στο Βέλγιο. Δηλαδή η ροή, αυτή η μεταναστευτική ροή δεν έχει μόνο επιπτώσεις για την παραμεθόρια χώρα. Ρωτώ λοιπόν, θα μπορούσαμε να έχουμε μία πιο οργανική και πιο ενιαία ή δυνατόν ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα αυτών. Διότι αυτό θα αποτελέσει και εγγύηση για ορισμένα ζητήματα. Δηλαδή όταν έχουμε τη Λιβύη και λέμε σήμερα η Ευρώπη πρέπει να πάει να τα βρει με τη Λιβύη και δεν μιλάμε για μια κύριε κροτσέτα σας παρακαλώ. Και όλα αυτά λοιπόν τα συζητάμε με την ε, Λιβύη, ξέροντας ότι η Λιβύη είναι μια χώρα που έχει πολλά άπλητα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. κυρία Μπαρζάκ. Λοιπόν, ε, λυπούμε και διαμαρτύρομαι γιατί οι δύο τοποθετήσεις που δεν ελήφθησαν υπόψη ε, ε, ήταν <coughs> τοποθετήσεις της ΓΚΟΕ. Λοιπόν, κύριε Διευθύντα, σίγουρα η Frontex είναι ένας τεχνικός οργανισμός. Αλλά ο τρόπος ο οποίος μας παρουσιάσατε τα πράγματα, ε, συγγνώμη για την έκφραση, είναι ένας τρόπος που πραγματικά μας παγώνει. Μιλάτε για λειτουργικότητα, για αποτελεσματικότητα, για καλύτερη χρήση των πιστώτεων. Η μόνη φορά που αναφέρεστε στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι στην πολιτική κατάρτιση των ε, συνοριακών φρουρών. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω δύο πράγματα. για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα στην Ευρώπη και για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τις χώρες τις οποίες έχει συμφωνίες η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Διευθυντά, δεν θεωρείτε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αρμόδιο και για αυτά τα θέματα. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις οποίες εσείς διαπιστώνετε και μετά τις καταγγέλλετε στα αρμόδια όργανα. Θα ήθελα να ξέρω επίσης ποιο, είναι το πρόγραμμα ε, κατάρτισης στα ανθρώπινα δικαιώματα. Μιλάτε επίσης για κακή χρήση της ε, υπηκότητας, μετά εκφράζεται ικανοποίηση για τις συλλήψεις. Και αυτό τι θέλει να πει, σε ποια βάση γίνονται αυτές οι συλλήψεις. Εκφράζεται ικανοποίηση για την ε, μείωση των παρανόμων ε, περασμάτων στα ευρωπαϊκά σύνορα, αλλά αυτό όμως γίνεται σε τρίτε, μέσω, στις τρίτες χώρες πια. Τι γίνεται με τη συνεργασία, λοιπόν πρέπει να τελειώνουμε. Θα τελειώνω, θα τελειώσω. Και αν δεν με διακόπτετε θα μιλήσω πιο, θα μιλήσω πιο γρήγορα. Λοιπόν, τι γίνεται με το Μαρόκο, με την Τινησία. Και τρίτο, ένας μετανάστης που θέλει να αμφισβητήσει την ηλιμένη θέση μπορεί να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του σχετικά. Σας ευχαριστώ. Διευθυντά έχετε το λόγο. Ευχαριστώ και πάλι. Δεν κατάλαβα την ερώτηση του κυρίου Έντσο για τις κοινέ έρευνε. Αν αφορούσε το κατά πόσον η Frontex θα έχει κοινέ ερευνητικέ ομάδε, η απάντηση είναι όχι. Δεν είναι η βασική μας δραστηριότητα. Θα ήθελα να, το, να μου διευκρινίσετε την ερώτηση αυτή που δεν την πολύ κατάλαβα, να σας πω την αλήθεια το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Είναι πολιτές πρόγραμμα και η Frontex παίζει σημαντικό ρόλο και στο πρόγραμμα και στις επιστροφές. Το πρόγραμμα Στοκχόλμης προσφέρει νέες δυνατότητες σχετικά. Επίσης, το γεγονός ότι τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας ενισχύει το ρόλο και την εικόνα ότι ο μεθοδιακός έλεγχος μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιο ανοιχτά για διάφορους στόχους όταν θεωρείται κατάλληλο. Αυτό είναι μια βασική προσέγγιση. Μπορούμε να δούμε ότι τα κράτη-μέλη καλούνται να είναι πιο δραστήρια. Η συμμετοχή είναι βασική αρχή του προγράμματος της Στοκχόλμης. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε υπομονετικοί, να έχουμε υπομονή. Ε, έχουμε μικρή διάρκεια της ε, ε, συνεργασίας του με αυτό, αλλά προχωράει. Το θέμα είναι, θέλουμε, είμαστε ικανοποιημένοι από την ταχύτητα ή θέλουμε πιο γρήγορες εξελίξεις. Κατόπιν. Αποφάσεις ό,τι αφορά την άρνηση εισόδου ή την σύλληψη παρανόμως ελχομένων λοδοπών. Να είμαι σαφής. Η Frontex δεν είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία που αποφασίζει την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πορεία του μετανάστη που συλλαμβάνουν οι μεθοριακοί φρουροί ε, μαζί με τις δραστηριότητές μας. Πάντα το κράτος μέλος είναι αυτό που θα κάνει την δραστηριότητα αυτή. Και οι αποφάσεις που αφορούν στη διαδικασία σύλλου στην σύλληψη, είναι αποφάσεις διοικητικού ή άλλης, διοικητικής ή άλλης φύσεως, είναι αποφάσεις, αποφάσεις της φιλοξενούσας χώρας. Δεν λέει η Frontex τι πρέπει να γίνει και τι πρέπει, ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί. Αυτό είναι σαφές. Και αυτό είναι ένα από τους λόγους για τους οποίους δεν είμαστε σε θέση να έχουμε να επηρεάσουμε τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν τα κράτη-μέλη. Εμείς προσπαθούμε να δώσουμε μια πιο μακρόπνοη εξέλιξη στην διαδικασία αυτή, χρησιμοποιώντας πιο ήπια εργαλεία, την κατάρτιση, τη συνεργασία, ε, αυτή είναι η προσέγγιση που ακολουθούμε. Το ίδιο ισχύει και με τις περιπτώσεις προσφύγων και με τα ζητήματα που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εδώ και δύο χρόνια έχουμε μια συμφωνία συνεργασίας και με την υπατιαρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και με τον ΔΟΜ η ύπατη αρμοστία εμπλέκεται συστηματικά στην διαμόρφωση των, ε, των ε, μαθημάτων κατάρτισης. Δυστυχώς δεν είμαι σε θέση να σας περιγράψω το περιεχόμενο των ε, μαθημάτων αυτών, αλλά αν θέλετε να σας τα στείλω αργότερα το ΓΙΟΝ η ύπατη αρμοστία έχει αξιωματικό σύνδεσμο που συνεργάζεται σε καθημερινή βάση, είναι αποσπασμένο σε εμά και συνεργάζεται σε καθημερινή βάση με τη Frontex. Και με το FRA, την υπηρεσία, ε, τον Οργανισμό για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Ε, τα παίρνουμε τα πράγματα αυτά πολύ σοβαρά και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προωθήσουμε πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων στον τομέα αυτό των ελέγχων στα σύνορα. Η ευρωπαϊκή πολιτική σε αυτή τη συμφωνία συνεργασίας. Νομίζω ότι είχαμε θετικές επιπτώσεις και από το γεγονός ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή επιχειρησιακή συμφωνία και με τις διμερείς συμφωνίες που έχουν κράτη-μέλη. Δεν είναι σημαντικό να κρίνουμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος. Το σημαντικό είναι ότι μπορούμε να συνεργαστούμε και να έχουμε επιχειρηματική συνεργασία με την τρίτη χώρα. Ωστόσο, οι προτεραιότητές μας είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τις τρίτες χώρες και να μην χρησιμοποιούμε για το σκοπό αυτό τα, τριτα κράτη-μέλη. Ελπίζω να κάλυψα όλες τις ε, πτυχές που τέθηκαν. Ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστώ Διευθυντά για τη σαφήνεια. Παρακαλώ να μείνετε εδώ, γιατί θα εξετάσουμε τώρα το τελευταίο σημείο που αφορά στο Frontex, είναι το έκτο, πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη συμπλήρωση του κώδικα συνόρων του Σέγγεν όσον αφορά την επιτήρηση των θαλασσίων εξωτερικών συνόρων στα πλαίσια της επιχειρησιακής συνεργασίας που συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα. Ο κύριος Μπούργος από το Συμβούλιο. Α, μετά την Κομισιόν. Στο Συμβούλιο, εμείς λάβαμε την πρόταση της Κομισιόν στις αρχές Δεκεμβρίου και ξεκινήσαμε τις εργασίες για να καταλήξουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα σε συμφωνία. Το χρονοδιάγραμμα είναι αρκετά σύντομο, είχαμε και επίσημες και ανεπίσημες ε, συνεδριάσεις. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε και ελπίζουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Είμαστε πάντως πεπισμένοι ότι δεν είναι κάτι το εύκολο. Ε, το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό για να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις σαν αυτές ε, που ακούσαμε σήμερα. Να σας θυμίσω ότι οι γενικές πολιτικές αρχές ε, ορίστηκαν στο 562 κάθετος 6 κανονισμό, ένα από τους πρώτους κανονισμούς που ελήφθησαν με συναπόφαση και εκεί ελήφθησαν τα πρώτα μέτρα για τα σύνορα. Είναι αποφάσεις λοιπόν κοινέ μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Ξέρουμε όμως ότι υπάρχουν πολιτικά προβλήματα που προκύπτουν ε, στο, ε, στα κράτη-μέλη. Υπάρχει και θέμα διεθνούς θαλασσίου δικαίου που πρέπει να εξετάσει το Συμβούλιο. Και υπάρχει και ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα, η αρχή του σεβασμού των ανθρωπίνων ε, ε, δικαιωμάτων και η μη επαναπρόθεση. Δεν είναι εύκολο να εργαστούμε. Ο χρόνος μας είναι πάρα πολύ ε, μικρός. Πάντως ε, πιστεύω ότι μπορούμε να σας στείλουμε ένα σχετικό έγγραφο ήδη αυτόν τον μήνα. Η Κομισιόν για να ολοκληρώσει την πληροφόρηση Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα για το υπόβαθρο της απόφασης. Οι επιχειρήσεις που περιέγραψε ο κ. Λάιτ είναι ιδιαίτερα στι θαλάσσιες επιχειρήσεις της Frontex. Λαμβάνουν ε, χώρα σε ένα περίπλοκο περιβάλλον με διεθνές δίκαιο, με ευρωπαϊκό δίκαιο, με πολλές ε, παρεκκλήσεις μεταξύ κρατών μελών σχετικά με την ερμηνεία των διατάξεων. Στόχος του σχεδίου απόφασης είναι λοιπόν πρώτον να καταστούν πιο αποτελεσματικέ οι κοινέ επιχειρήσει που συντονίζει η Frontex. Δεύτερον, υπάρξει ένα σαφέστερο προβλέψιμο νομικό πλαίσιο που θα επιτρέπει πλήρη συμμετοχή στα κράτη-μέλη. Και τρίτον, πολύ σημαντικό και αυτό, να υπάρξει πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και συμπεριλαμβανομένη και τη αρχή τη μη επαναπροώθηση τη επιχειρήση τη Frontex. Αυτό είναι πολύ τεχνικό θέμα. Η απόφαση μπαίνει σε λεπτομέρειες σχετικά με το πώς οι επιμέρους διοικητές, οι αξιωματικοί θα πρέπει να δρουν, τι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όταν λαμβάνουν αποφάσεις στη θάλασσα ε, μεσουσών των επιχειρήσεων. Επίσης είναι και θέμα ερμηνείας η απόφαση αυτή. Θα πρέπει να υπάρξουν κοινέ κατευθυντηρίε γραμμέ, μια κοινή άποψη σχετικά με το διεθνέ δίκαιο και το ευρωπαϊκό δίκαιο και πώ θα πρέπει να εφαρμόζονται αυτά από τα κράτη-μέλη όταν συνεργάζονται στα πλαίσια επιχειρήσεων τη Frontex. Γι' αυτό έλαβε την απόφαση ο Αντιπρόεδρος Μπαρό να προετοιμάσει το σχέδιο απόφασης της Κομισιόν ε, στα πλαίσια του κώδικα των συνόρων και την μεταβίβαση των ε, αρμοδιοτήτων που προεβλέπεται ήδη στον κώδικα αυτό για τα σύνορα και να δημιουργηθούν έτσι οι ευρωπαϊκοί κανόνες για την ε, πραγματοποίηση των κοινών επιχειρήσεων της Frontex. Ε, συνεργαστήκαμε πολύ με τα κράτη-μέλη, είναι περίπλοκο το θέμα και έπρεπε να προσπαθήσουμε πολύ, ούτως ώστε να έχουμε κοινή κατανόηση των σχετικών κανόνων. Με, ε, ένα πρώτο σχέδιο παρουσιάστηκε στην Επιτροπή τον Φεβρουάριο μετά έγιναν πολλές ε, θεωρήσεις και η τελευταία εκδοχή του υπευλήθη στην Επιτροπή των Συνόρων Οκτώβριο ε, υπήρχαν 7 ψήφοι κατά και αποχές, πράγμα που δεν επέτρεψε να καταλήξει η Επιτροπή σε γνωμοδότηση ε, ούτε υπέρ ούτε κατά. Ε, ακόμα δίστανται λοιπόν οι απόψεις, κυρίως επί της νομικής βάσεως και θέματα διάσωσης, που θα πρέπει να συμπεριληφθούν ή όχι. Κάποια κράτη-μέλη θα προτιμούσαν μη δεσμευτικέ κατευθυντήριες γραμμές, Υπάρχουν διαφορές απόψεων και σε σχέση με τη διαφορετική ερμηνεία του διεθνούς δικαίου που αν θέλετε είναι ε, η βάση όλων αυτών και γι' αυτό υποβάλαμε και το σχετικό σχέδιο απόφασης και τέλος θα πρέπει ίσως να αναδειχθούν και διαφορετικές απόψεις μεταξύ κρατών μελών σχετικά με τον ορισμό του κανόνα της ε, αποβίβασης μετά από διάσωση ή μετά από σύλληψη ή αναχέτηση. Επειδή λοιπόν δεν υπήρξε γνωμοδότηση από την Επιτροπή του Κώδικα των Συνόρων, η Κομισιόν υποχρεώθηκε να υποβάλει πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου και αυτό τώρα το χειρίζεται το Συμβούλιο, όπως είπε και ο κύριος Μπούργος. Με... Η προθεσμία είναι τώρα 7 Φεβρουαρίου για το Συμβούλιο και 7 Απριλίου για το Κοινοβούλιο να ασκήσει το δικαίωμα κοινοβουλευτικού ελέγχου το τελευταίο. Είμαι στη διάθεση της Επιτροπής, κύριε Πρόεδρε, για τυχόν συμπληρωματικές ή άλλες ερωτήσεις επί του θέματος. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπουσουτήλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις, ε, όχι δύο παρατηρήσεις θα κάνω. Το πρώτο διαδικαστικό. Δεν κατάλαβα πολύ καλά Ποια είναι η νομική βάση αυτής της πρωτοβουλίας, γιατί αν κατάλαβα καλά εδώ λειτουργούμε στα πλαίσια των κανόνων της επιτροπολογίας. Θα ήθελα όμως οι νομικές υπηρεσίες, αν εκπροσωπούνται σήμερα, να μας πούν ποια ακριβώς είναι η νομική μας βάση εδώ και ποια είναι τα προνόμια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, επί του θέματος του συγκεκριμένου. Ε, και εις επίμετρον, η συνθήκη της Λισαβόνας επηρέασε την πρωτοβουλία αυτή που νομίζω ότι αρχικά υπευλήθη πριν από τη Λισαβόνα, ενώ η απόφαση θα ληφθεί μετά τη Λισαβόνα. Ναι, Ε, ε λοιπόν, νομικές, ε, νομική βάση. Αν οι νομικές υπηρεσίες δεν μπορούν να μας πούν σήμερα, μπορούμε να τους απευθύνουμε γραπτό στο αίτημα και θα απαντήσουν και εκείνοι γραπτός. Δεύτερο πολιτικής μάλλον φύσεως ε, παρατήρηση ε, θέμα. Εδώ έχουμε ένα, μια τεχνική πρωτοβουλία ή μια πρωτοβουλία που φαίνεται να είναι τεχνικής φύσεως ενώ στην πραγματικότητα έχει τεράστια πολιτική σημασία. Πρέπει λοιπόν, θεωρώ, να σκεφτούμε πολύ προσεκτικά τις πολιτικές επιπτώσεις της πρωτοβουλίας αυτής. Ειδικότερα, η ερώτησή μου είναι η εξής. Στο Κοινοβούλιο αυτό επανειλημμένα έχουμε δηλώσει ότι είναι πολύ σημαντική η αλληλεγγύη, ο επιμερισμός των βαρών και η ετοιμότητα των κρατών μελών από κοινού να αναλαμβάνουν την ευθύνη όταν πρέπει να αντιμετωπίσουν την εισρωή των μεταναστών. Αν αντιλαμβάνομαι ορθώς, εδώ έχουμε μια απόφαση του Συμβουλίου που αποφασίζει ότι μια συγκεκριμένη χώρα είτε θα είναι η χώρα Α, η Β, η Γ, μια χώρα θα πρέπει να επιλαμβάνεται όσων εισέρχονται στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Αυτό είναι σε σαφή αντίφαση ε, με τις αρχές του Κοινοβουλίου που τάσεται υπέρ της ελληνικής, ενώ το Συμβουλίο μας λέει όχι. Αλληλεγγύη δεν έχει. Μία χώρα θα πρέπει να δέχεται την, ε, το ρεύμα αυτό, την εισρωή αυτή. Νομίζω ότι αυτό για το κοινοβούλιο μας δεν είναι αποδεκτό. Κάθε άλλο. Γι' αυτό πρέπει να δούμε πολύ προσεκτικά τις προνομίες μας πριν καταλήξουμε σε τυχόν συμπεράσματα για το θέμα. Ευχαριστώ. Η κυρία Φλότσχα. Πιστεύω ότι είναι καλή και ευχθέα η παρουσίαση που έγινε διότι όταν θέλουμε εμείς να συντονίσουμε το, το Frontex θα πρέπει να διασφαλίσουμε επίσης ότι και τα κράτη-μέλη σέβονται όλους τους νόμους και κανόνες. Πρόκειται λοιπόν για κάτι το απαραίτητο, το κατεπήγον. Ερώτηση. Μετά από την παρουσίαση του διευθυντή του Frontex, ο οποίος αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη και αρμοδιότητα για αυτά τα θέματα, σίγουρα ε, παραλύουν έτσι οι εφαρμογές αυτές των, των κατευθυντηρίων γραμμών. Επίσης, ε, σύμφωνα με τις διάφορες συμβάσεις, είναι ιδιαίτερα ενοχλητικό όταν λέμε ότι θα πρέπει να κατανέμονται κατά προτεραιότητα ή πρόσφυγες ε, στην ε, χώρα ε, από την οποία προέρχονται. Αλλά αυτό παραβιάζει όλους τους κανόνες που έχουμε και για τα δικαιώματα των προσφύγων αλλά και για το θαλάσσιο το Διεθνές Θαλάσσιο Δίκαιο που λέει ότι όταν βοηθάμε ναυαγούς το, πιο, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να τους πάμε στην πιο ασφαλή και κοντινή στεριά. και δεν μπορούμε εμείς ε, χρησιμοποιώντας ε, ένα ε, υπεφεύγοντες όρους να κρύβουμε πίσω από το δάχτυλό μας την ανομοιογένεια του δικαίου χορήγησης ασύλου που ισχύει στα κράτη-μέλη. Ο Μωράες. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συμφωνώ με τους προηγούμενους ομιλητές είναι ένα θέμα πολύ σύνθετο και με σοβαρές πολιτικές συνέπειες. Μία από αυτές είναι ότι το άρθρο 4 της πρότασης της Επιτροπής περιγράφει, περιλαμβάνει μια κατάσταση που στο κείμενο του Συμβουλίου ε, μιλά για μια επαναπροώθηση και άλλες, δομές προστα... και άλλες μορφές προστασίας του πρόσφυγα, χωρίς ωστόσο να αναφέρεται ρητά το κείμενο αυτό υπάρχει πραγματική πιθανότητα εφαρμογή, ε, υλοποίησης, επαναπροώθησης. Αυτό το, το ζήτημα το, το ανέφεραν πολλές ΜΚΟ. Θε, άλλο ζήτημα, επιτροπολογία. Ε, με βάση, μετά την θέση ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, τι ρόλο έχει το Κοινοβούλιο στη διαδικασία αυτή. Μπορεί να μην μπορείτε να απαντήσετε, αλλά εγώ, αν κατάλαβα καλά, το Κοινοβούλιο έχει τη δυνατότητα να εξετάσει το κείμενο στη δική μας επιτροπή δύο μήνες μετά. Δεν ξέρω ποιο ρόλο ακριβώς έχει το Κοινοβούλιο, ξέρω ότι είναι περίπλοκο ο ρόλος αυτός, αλλά νομίζω ότι έχουμε μια τέτοια δυνατότητα με βάση τη Λισαβόνα. Σωστά αναφέρει και είπε και ο κύριος Μπουσούτελ και η κυρία Φιλότρο ότι αυτό το κείμενο έχει ε, πολύ μεγαλύτερες πολιτικές συνέπειες από αυτές που νομίζουμε. Η κύριε Χένις Πλασκάρ για τη νομική βάση καλό θα ήταν να ακούσουμε και την άποψη του Συμβουλίου που και εκεί παρεύουν για το, για το θέμα αυτό. Αύριο το πρωί υπάρχει μια συνάντηση των νηστών και θα ήταν σκόπιμο να έχουμε μπροστά μας αύριο το πρωί την νομική γνώμη πριν τη συνάντηση των συντονιστών. Το Κοινοβούλιο μπορεί ε, να πει ναι ή όχι μόνο αν κατάλαβα καλά, αλλά πρόκειται για σημαντική συμφωνία. Συμφωνώ επίσης απόλυτα με τις ανησυχίες του Σάιμον σε ό,τι αφορά την κατανομή των βάρων των πέντε sharing, αλλά ούτως ή άλλως αυτό θα είναι καθηγητήρες γραμμές για την εφαρμογή του burden sharing, γιατί κάποια κρατημέλη δεν είναι δεν θέλουν να μετάσχουν στο burden sharing γιατί δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία οι διαδικασίες. Μην ξεχνάτε ότι το Frontex άρχισε να λειτουργεί το Νοέμβριο του 5. Τώρα είμαστε εν έτη 2010 και ακόμα περιμένουμε αυτές τις καθηγητήριες γραμμές. Χρόνια και χρόνια συζητάμε. Αν θα, ενώ για το θέμα αυτό, ενώ κανονικά θα πριν κάνει λειτουργήσει το Frontex έπρεπε να υπάρχουν οι καθηγητήριες γραμμές γιατί αυτό θα έχει αποφύγει πολλά προβλήματα. Και πολλές φορές η Επιτροπή έκανε ότι, και η Επιτροπή έκανε ότι μπορούσε για να το προωθήσει τα κράτη-μέλη, αλλά τα κράτη-μέλη δεν το ήθελαν. Εν τέλει, ωστόσο πιστεύω, γιατί αυτό κατάλαβα, υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα πρέπει να λυθεί μεταξύ Μάλτα και Ιταλίας. Θα εκτιμούσε ωστόσο να μπορούσε το Συμβούλιο να παρέμβει στην διαμάχη αυτή ούτω ώστε να ξέρουμε πώς το που κατευθυνόμαστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ορισμένες από τις παρατηρήσεις του κυρίου Μπουσοτήλ εμπλέκουν τις νομικές υπηρεσίες και ίσως ε, χρειαστεί να δοθεί γραπτή απάντηση. Δεν ξέρω αν η νομική υπηρεσία στο μεταξύ μπορεί να βοηθήσει. Και μετά θα δώσω το λόγο στο Διευθυντή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω μια σύντομη παρέμβαση σε αυτό το σημείο. Με κάθε μετριοπάθεια ευχαριστώ την Κομισιόν και το Συμβούλιο για το έργο τους σε αυτό το σημαντικό θέμα. Νομίζω ότι διευκρινίστηκε στην Επιτροπή εδώ και ε, στα πλαίσια της συζήτησης ότι αν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν μπορούν να συμφωνήσουν αυτό σχετικά με τα μέσα, αυτό είναι πρόβλημα για μας. Και για μένα ήταν πρόβλημα εδώ και χρόνια. Αυτά τα προβλήματα τα βλέπω εγώ ξανά και ξανά. Δουλειά μου είναι να προβλέψω σωστή λειτουργία των επιχειρήσεων. Δεν θα μπω εγώ στα πολιτικά θέματα που ανέκυψαν. Οπότε η έκκλησή μου είναι να βρεθεί λύση ούτως ώστε να προχωρήσει το μέσον αυτό, ε, βεβαίως στο σωστό φόρουμ με τη σωστή νομική βάση και πολύ καλό θα είναι να έχω και εγώ κάποιες οδηγίες ε, έγκυρες για να μπορώ και να μπορούμε όλοι μας στη Frontex να δουλεύουμε. Εγώ ουσιαστικά έδωσα το λόγο βέβαια στις νομικές υπηρεσίες δεν ξέρω αν η νομική υπηρεσία μπορεί να συνεισφέρει ή θέλει να τα δώσει γραπτός μετά. Ε, κοιτάστε, εμείς ε, καταγράψαμε την ερώτηση του κυρίου Μπουσουτήλ. Ξέρετε ότι τα θέματα επιτροπολογίας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα. Μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας, η παλιά απόφαση του 99 όπως τροποποιήθηκε το 2006 για την επιτροπολογία έχει πεθάνει. Δεν χρησιμοποιείται πλέον, αλλά όλες οι νομοθετικές πράξεις που εγκρίθηκαν πριν από τη θέση σε ισχύ της Λισαβόνας υπό το καθεστώς της επιτροπολογίας που ανέφερα παραμένουνε διότι αποτελούν κομμάτι του κοινοτικού κεκτημένου. Οπότε όλες οι αποφάσεις επιτροπολογίας που τέθησαν σε ισχύ ε, πριν από τη Λισαβόνα παραμένουν. Μία επιτροπή λοιπόν που συστάθηκε πριν από τη συνθήκη της Λισαβόνα θα συνεχίσει να, ε, την πορεία της όσο η βασική ιδρυτική της πράξη ισχύει. Σε περίπτωση που αλλάξει η ιδρυτική της βάση, τότε ό,τι τροποποίηση γίνει θα γίνει βάση της Λισαβόνας, η οποία στο άρθρο 291 προβλέπει ότι η παλιά απόφαση που ονομάζουμε επιτροπολογία θα πρέπει να αντικατασταθεί από έναν κανονισμό που θα αποφασίζεται σε συναπόφαση μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου κατόπιν υποβολής προτάσεως της Κομισιόν. Και η Κομισιόν μας είπε ότι θα κοιτάξει να παρουσιάσει τις ε, προτάσεις της το συντομότερο δυνατόν. Αυτά γενικά για την παλιά απόφαση σχετική με την επιτροπολογία. Τώρα με την δική μας συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να εξετάσουμε το σχετικό έγγραφο διότι θα πρέπει να δούμε αν αυτό το μέτρο βασίζεται στην παλιά απόφαση της επιτροπολογίας οπότε εδώ πρόκειται απλά και μόνο για εφαρμογή ή αν πρόκειται για αλλαγή. Και τότε αν είναι αλλαγή πρέπει να αλλάξουμε κεφάλαιο και να μεταφερθούμε στη Λισαβόνα. Ζητώ όμως να μου δώσετε μία περίοδο χάριτος και να απαντήσω γραπτός στην ερώτηση που θα μου στείλει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Φυσικά και θα σας στείλουμε μία γραπτή ερώτηση. Είναι ανοιχτό λοιπόν το θέμα. Οπότε επειδή έχουμε καθυστερήσει λέω να αρχίσουμε να ψηφίζουμε αν συμφωνείτε φυσικά. Ψηφίζουμε το σημείο 8 απαλλαγή για το 2008 η συγητής Λόπες Αγγιλάρ Είμαστε έτοιμοι. Ξέχασα την ε, κάρτα μου. Μπορώ να ψηφίσω σηκώνοντας το χέρι, διανατάσεις της χειρός. Quindi per chi non ha la tessera, il tesserino, la levata di mano dovrebbe essere Ναι, εντάξει, όταν ε, δεν έχει κανείς την ηλεκτρονική κάρτα, τότε η άρση της χειρός ε, είναι ισοδυναμή. Σημείο 8. Τροπολογία του Μπουσουτήλ. Ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Σημείο 9 έχουμε δύο τροπολογίες, ψηφίζουμε. Την πρώτη τροπολογία της κυρίας Βερζή, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερη τροπολογία, Μπουσουτήλ. Με την προφορική τροπολογία, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται τελική ψηφοφορία. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σημείο, σημείο 10 και εδώ έχουμε μία τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Επόμενο σημείο. Και εδώ δύο τροπολογίες. Ψηφίζουμε την πρώτη τροπολογία της κυρίας Μπερσά. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 2 Μπουσουτήλ με την προφορική αλλαγή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Για την Τσέπολ τρεις τροπολογίες. περ της πρώτης τροπολογίας κυρίες Βερζά. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερη τροπολογία πάντα της κυρίες Βερζά. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτη τροπολογία με την προφορική τροπολογία που σου θέλει, Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Frontex. Τροπολογία του Μπουσουτήλ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η δεύτερη αποσύρεται, η τρία γίνεται δύο του κυρίου Μπουσουτήλ, πάντα με την προφορική αλλαγή, υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Λοιπόν, τελικό κείμενο, υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Κοέλιο που ήρθε στο μεταξύ. Το σημείο 7 λοιπόν μπορούμε να το, να το ξεκινήσουμε και να το παρουσιάσει. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά τις θεωρήσεις ε, μακράς διάρκειας υπάρχουν δύο εκθέσεις. Ε, ήταν υποχρεωτικό να γίνει αυτό, διότι πριν την συνθήκη της Λισαβόνας ήταν, ε, κάποια θέματα, υπήρχαν κάποια θέματα που υπάρχονταν στη συναπόφαση, ενώ κάποια άλλα που υπάρχονταν στην διαβούλευση. Μετά τη θέση ισχύ της ε, Λισαβόνας υπάρχει συναπόφαση σε όλους τους τομείς που αφορούν τις δύο εκθέσεις η Σουηδική Προεδρία είχε προτείνει να δουλέψουμε με ένα κείμενο και όχι με δύο. Η πρότασή μου λοιπόν είναι να ακούσουμε την θέση της ε, Ισπανικής Προεδρίας και αν θέλει να λάβει θέση και η Κομισιόν να ακούσουμε και αυτή. Κατόπιν να μιλήσω εγώ έχοντας ακούσει το Συμβούλιο και την Επιτροπή πάνω στο κείμενο. Ωραία. Η Ισπανική Προεδρία παρακαλώ. Κύριε Μπούργος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Την ουσία του θέματος την εξήγησε ο κύριος Κοέλιο. Μετά τη θέση ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας χρειάζεται να αναμορφωθεί ο τρόπος παρουσίασης των δύο πρωτοβουλειών. Είμαστε σε επαφή με τον εισηγητή και συμφωνούμε να προχωρήσουμε με τον τρόπο που ανέφερε ο ίδιος, ένα κοινό δηλαδή ψήφισμα. Με, τις, ε, με βάση τις επαφές που είχαμε πιστεύουμε ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Κοινοβούλιο στον τομέα αυτό. Ε, μπορούμε να συζητήσουμε την ΑΒ τοπολογία, αλλά επί της ουσίας νομίζω ότι υπάρχει μια συμφωνία που μπορεί να προχωρήσει γρήγορα σχετικά. Ευχαριστώ η Επιτροπή. Θα είμαι πολύ σύντομη. Επιβεβαιώνουμε αυτά που είπε ο κύριος Κοέλιο. Ο λόγος τον οποίο υποβάλαμε δύο προτάσεις πέρσι ήταν ότι θέματα που κάλυπτε η πρόταση υπάγονταν στη διαδικασία συναπόφασης. Άλλοι τομείς, ωστόσο, είχαν παραμείνει στη διαδικασία της συναπόφασης. Μετά τη θέση ισχύ της Λισαβόνα, της συνθήκη δηλαδή της Λισαβόνα. όλη η πρόταση είναι πλέον βάση της διαδικασία συναπόφασης. Δεν δικαιολογείται λοιπόν να έχουμε δύο χωρίστες προτάσεις, γι' αυτό συμφωνούμε με το Συμβούλιο την Ισπανική Προεδρία να συγχωνευτούν οι δύο προτάσεις. Ευχαριστώ. Θέλει να λάβει ξανά το λόγο ο κύριος Κοέγιο. Ευχαριστώ. Ήθελα πριν να σας πω ότι κατά την άποψή μου πρόκειται για μια τεχνική τροπολογία που έχει ωστόσο το πλεονέκτημα να καταστεί σαφέστερη την διαδικασία παρέμβαση του Κοινοβουλίου. Προτείνω σε όλους τους συναδέλφους να δεχθούμε τη διαδικασία, τη συγχώνευση δηλαδή των δύο εκθέσεων, να ευχαριστήσω τη Γραμματεία της Επιτροπής που ήδη προετοίμασε τη συγχώνευση του διατακτικού των δύο κειμένων και να ζητήσω ε, η δουλειά αυτή, το κείμενο αυτό να αποστελεί ήδη σήμερα σε όλους τους συναδέλφους της Επιτροπής μας. Είχαμε προβλέψει ως προθεσμία υποβολή τροπολογιών τη 18η Ιανουαρίου. Σε μια εβδομάδα δηλαδή. Οι συνάδελφοι που είχαν ετοιμάσει τροπολογίες θα μπορέσουν ευκολότερα να ετοιμάσουν τις τροπολογίες με ενοποιημένο το κείμενο και όχι με δύο εκθέσεις ξέχωρα. Αν είχαμε λοιπόν τη δυνατότητα να δούμε το κείμενο, το ενοποιημένο κείμενο τώρα θα ήταν ευκολότερο να υποβάλουν εμπρόθεσμα τις τροπολογίες συνάδελφοι και να συμβαστούμε το χρονοδιάγραμμα που έχουμε υιοθετήσει. Με το ενοποιημένο κείμενο όπως προτείνει η Ισπανική Προεδρία θέλω να τονίσω και κάποιοι ήδη το είδαν ότι βάσει του κανονισμού ε, άρθρο 37 χρειάζεται να υπάρξει διαβούλευση με την νομική επιτροπή, με την Επιτροπή Νομικών υποθέσεων όταν υπάρχει τροπολογική της νομικής βάσης. Αυτό ωστόσο μπορεί να γίνει χωρίς να φοβόμαστε λόγω να έχουμε προβλήματα λόγω χρονοδιαγράμματος. Αν συμφωνεί η Επιτροπή με την πρόταση που έχει υποβάλει ο συνάδελφος Κοέλιο να προχωρήσουμε. Παρακαλώ. Δεν βλέπω κανέναν από την Επιτροπή μας να θέλει να λάβει το λόγο. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 18 Ιανουαρίου για το ενοποιημένο κείμενο. Συμφωνούμε όλοι. Ωραία κύριε Κορέγιο, προχωρούμε. Δικαίωμα διερμηνίας και μετάφρασης σε ποινικέ διαδικασίες, σε ποινικέ δίκες δηλαδή. Η Βαρόνι Λάτφορντ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως γνωρίζετε, η πρόταση που εισηγήθηκα οδήγησε σε έκθεση και στηρίχθηκε σε έκθεση το προηγούμενο Οκτώβριο. Κατέπεσε λόγω της συνθήκης της Λισαβόνας, άρα πρέπει να αρχίσει στα πλαίσια της Λισαπόνας νέα διαδικασία για πρόταση οδηγίας γιατί η έκθεσή μου δεν ψηφίστηκε ούτε στην Επιτροπή, ούτε στην Ολομέλεια, αφού δεν είχε λήξει, δεν είχε παρέλθει το χρονοδιάγραμμα. Άρα λοιπόν, τώρα μπαίνουμε στο πλαίσιο της ε, συνομοθεσίας με το Συμβούλιο το Συμβούλιο την τελευταία μέρα πριν από τη Λισαβόνα, 30 Νοεμβρίου δηλαδή, ενέκρινε ε, ψήφισμα για έναν οδικό χάρτη, χάρτη πορείας για σταδιακή προσέγγιση αυτών των ε, δικονομικών δικαιωμάτων, οπότε αυτό είναι ένα ειδικό μέτρο στα πλαίσια του οδικού χάρτη. Χαίρομαι πολύ που συνεχίζομαι την ε, καλή πορεία μας και καλές εργασίες μας σε αυτό το μέτρο διερμηνίας και μετάφρασης. Εγώ συνήθως δεν υποστηρίζω τις πρωτοβουλίες των κρατών μελών με τόσο ενθουσιασμό, αλλά είναι ο ταχύτερος τρόπος για να ε, επιτελεστεί πρόοδος λόγω της ε, μεσοβασιλείας αυτής, αν θέλετε, που σημειώθηκε και τα εμπόδια που ίσως θα καθιστούσαν αναγκαία νέα ε, αξιολόγηση επιπτώσεων που θα έπαιρνε κανένα εξάμεινο. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει ο ικανός αριθμός των κρατών μελών, των βουλευτών με συγχωρείτε, 27 νομίζω, που αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αυτή τη διαδικασία. Ε, είχαμε βέβαια από το περασμένο καλοκαίρι και την αξιολόγηση επιπτώσεων της Κομισιόν. Οπότε είναι μια διαδικασία χρήσιμη, ρεαλιστική, που έτσι όπως είναι τα πράγματα μας επιτρέπει να μην καθυστερήσουμε και να μην υπάρξει στασιμότητα στη διαδικασία. Και μάλιστα ε, είναι στόχος εφικτός η συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση, ούτως ώστε όλα αυτά να τα ολοκληρώσουμε επί Ισπανικής Προεδρίας. Τώρα, σε συμφωνία με τους χειώδεις από τις άλλες ε, ομάδες υπέβαλα δύο προφορικές ερωτήσεις που ελπίζω να διατηρηθούν στην ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας την επόμενη εβδομάδα. Αντίθετα με κάποιες φήμες, ε, δεν προτίθεμαι να αποσύρω αυτές τις προφορικές ερωτήσεις. Είναι αλήθεια ότι η διατύπωση ε, τώρα είναι λίγο ξεπερασμένη, γιατί η διατύπωση ε, ήταν της 1 η Δεκεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία δεν ξέραμε τι τροπή θα παίρνανε τα πράγματα. Δεν αξίζει τον κόπο να ξανασυντάξουμε τις ερωτήσεις, αλλά επειδή υπάρχει δυνατότητα, καλό είναι να γίνει συζήτηση, υπάρχει χώρος. Το σημαντικό ιδιαίτερα στα πλαίσια της Νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της κατάρτισης του προγράμματος δράσης για την υλοποίηση του προγράμματος της ε, Στοκχόλμης είναι να είμαστε εστιασμένοι όλοι, επικεντρωμένοι και να υπάρξει και μια πολιτική δέσμευση εις ό,τι αφορά τη συνέχιση της προόδου για την υλοποίηση του οδικού χάρτη. Και αυτό το μέτρο είναι ένα πρώτο βήμα. Πρώτο ανάμεσα σε άλλα προβλεπόμενα. Εγώ είμαι πεπισμένη ότι όλα στον οδικό χάρτη και άλλα ακόμα όχι μόνο χρειάζονται, αλλά έχουν καθυστερήσει και πολύ. Το Κοινοβούλιο πάντα ήθελε ένα συνολικό μέτρο. Εμεί θέλαμε μια διαδικασία. είτε οδηγία ή κάποιο άλλο νομοθέτημα. Δεν ε, τα καταφέραμε λόγω της πολιτικής πραγματικότητας που υπήρχε. Όπως και αν βλέπουμε το ποτήρι, μισοάδιο ή μισογεμάτο, πρέπει να προσπαθήσουμε να μεγιστοποιήσουμε το περιεχόμενο και την ταχύτητα με την οποία κινούμεθα σε αυτά τα θέματα. Δεν θα μακρηγορήσω. Ε, παρουσιάζοντας προσωπικές εμπειρίες, αλλά χειρίζομαι διάφορες τέτοιες υποθέσεις ε, αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, όπου στην δική μου εκλογική περιφέρεια υπάρχει υποστήριξη, υποδοκιμή σοβαρή όμως, γιατί στην εκλογική μου ε, περιφέρεια υπήρχαν περιστατικά ε, όπου θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία με άλλες χώρες. Χρειάζεται λοιπόν συνεργασία, ούτως ώστε να μας υποστηρίξει και ο κόσμος όταν μιλάμε για ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και αμοιβαία αναγνώριση κλπ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι ένα κομμάτι της αμοιβαία εμπιστοσύνη που χρειάζεται, που χρειαζόμαστε και που δεν υπάρχει. Κινούμεθα σε στρώμα λεπτό πάγου εδώ. Πρέπει λοιπόν να γίνουν οι διαπραγματεύσεις, να λυθούν όλα αυτά μέσα στις διαπραγματεύσεις και υπάρχουν και ορισμένα θέματα που θα τα δείτε και σε σχέση με το κείμενο του Συμβουλίου 23 Οκτωβρίου Ακανθόδη θέματα προς επίλυση εις ό,τι αφορά το εύρος των δικαιωμάτων που ε, διασφαλίζονται υπό την προτινωμένη οδηγία. Αυτό που θέλω να σημειώσω είναι ε, η δέσμευση, να βεβαιωθούμε ότι θα ευθυγραμμιστούμε με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη σχετική νομολογία, ούτω ώστε να υπάρχει ε, συνάφεια μεταξύ συστήματος Τρασβουργού και Λουξεμβούργου, αν θέλετε, ακόμα και αν υπάρχουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης λεπτομερέστερα δικαιώματα. Τα κοινά δεν πρέπει να παρεκκλίνουν ως προς την ερμηνεία τους, αλλιώς θα δυσκολευτούμε πολύ. Και χαιρετίζω πολύ την υποστήριξη και το feedback, την ανάδραση από το Συμβούλιο της Ευρώπης που θεωρώ ότι είναι χρησιμότατο. Τέλος να πω ότι προβλεπόταν με την απόφαση πλαίσιο να συνοδεύσω με το νομικό μέσο, το νομοθετικό μέσο με ψήφισμα. Όχι το ψήφισμα για τον οδικό χάρτη, άλλο είναι αυτό. ψήφισμα για την ερμηνεία, για τη διερμηνία και την μετάφραση. Και να είναι, αν θέλετε, μη δεσμευτικό δίκαιο. Αυτό που τα κράτη-μέλη θέλουν να είναι δεσμευτικό δίκαιο. Τώρα, εγώ θα προέτεινα, θα έλεγα ότι θα πρέπει να συνεργαστεί ο συνομοθέτη στο Κοινοβούλιο και στο ψήφισμα, όχι μόνο στην οδηγία. Πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε από τι νομικέ υπηρεσίε μα να αποφανθούν σχετικά με το αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, αν θα έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι το, η ιδεολογική έκθεση του Συμβουλίου ε, εμέσως αναφέρει ότι δεν πρέπει να συμμετάσχουμε εμείς. Αξίζει τον κόπο μας να το δούμε, γιατί πώς θα αποφασίσουμε το νομοθέτημα, την οδηγία, αν δεν ε, δούμε τι θα αναφέρει το ψήφισμα, το οποίο είναι συμβουλευτικό. Και δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε την οδηγία αν δεν ξέρουμε τι θα λέει το ψήφισμα. Ζητώ λοιπόν οι νομικές υπηρεσίες να το δουν αυτό το ζήτημα και να γνωμοδοτήσουν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αγγιλέρα από την Ισπανική Προεδρία τώρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω να ευχαριστήσω για την Προεδρία, για την ε, ευκαιρία που μου δίνεται να παρουσιάσω την πρωτοβουλία αυτή που την υπέβαλαν 13 κράτη-μέλη για την έγκριση της οδηγίας για τα δικαιώματα διερμηνίας και μετάφραση σε ποινικέ δίκες. Το περιεχόμενο της ε, πρωτοβουλίας αυτής περιλαμβάνει κατά βάση το κείμενο που συζητήθηκε στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων τον Οκτώβριο του 2009 και που στηρίχθηκε σε μια πρόταση που είχε υποβάλει τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου η Επιτροπή. Ο στόχο ε, που επεδίωκαν τα κράτη-μέλη, τα 13 κράτη-μέλη που ανέλαβαν την πρωτοβουλία αυτή, ήταν να διευκολύνει την συνέχιση της διαδικασίας αυτής που είχε ξεκινήσει στο προγενέστερο εξάμεινο και για το οποίο τουλάχιστον στο Συμβούλιο υπήρχε σημαντική πρόοδος. Ο στόχος λοιπόν ήταν να εκμεταλλευτούμε και την θετική συγκυρία και που είχε πραγματοποιηθεί και να αποφύγουμε καθυστερήσεις που θα συνέπιπταν από τις αλλαγές λόγω της θέσης ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας και της εκλογής της Νέας Επιτροπής. Ωστόσο, οι περιστάσεις οδήγησαν στο να είναι το κείμενο αυτό η πρώτη πρόταση που υπάγεται στη στην απόφαση στα πλαίσια της δικαστικής και ποινική συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό θέλω να τονίσω ότι η Ισπανική Προεδρία είναι απόλυτα ε, πρόθυμη να συνεργαστεί σε στενή, στενά με το Κοινοβούλιο και να πετύχει μια ικανοποιητική συμφωνία το ταχύτερο δυνατό. Ε, όπω είπε και η κυρία Άλφοντ, ή δυνατόν σε πρώτη ανάγνωση και όπως και ανέφερε η κυρία αναγνωση και όπω επίσης, η κυρια αλφοντ επίση, η πρώτη αυτη δεν σταματά εδώ. Είναι το πρώτο βήμα για ένα ευρύτερο πρόγραμμα που έχει στόχο την προσέγγιση τη νομοθεσία για τις εγγύσεις που υπάρχουν στις ποινικέ δίκες και που θα συνεχίσουν να τηρούν το νοδικό χάρτη του 2009 και θα καθετευθύνουν τις εργασίες της Επιτροπής. Επίσης, σε σχέση με αυτό που είπε η κυρία Λάντφορντ ε, στην τελευταία παρατήρησή της είναι ότι η πρόταση της Προεδρίας η πρόταση αυτή κατά την άποψη της Προεδρίας επεκτείνεται και σε μια πρόταση απόφαση του Συμβουλίου και 100 Μερών για, τα, για μέτρα που θα ε, υλοποιήσουν στην πράξη τα συγκεκριμένα μέτρα, παρότι δεν υπάρχει το ίδιο το κείμενο στη διαδικασία συναπόφαση. Το περιεχόμενο της απόφασης αυτή που συνδέεται πάρα πολύ στενά με την οδηγία και δεν θα είχε νόημα να αποκλίνουν μεταξύ του, θα έπρεπε και αυτή να ακολουθεί τον ίδιο δρόμο όπως σας είπα, τη διάθεση που προανέφερα την επεκτείνουμε και στο σημείο αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή τώρα έχει το λόγο. Η κυρία Κάρολιν Μόργαν. Ευχαριστώ. Thank you very much. I would like... Ευχαριστώ πολύ. Πέντε σύντομες παρατηρήσεις. Πρώτον, η Κομισιόν χαίρεται που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2009 η πρόταση θεωρούμε όπως το Κοινοβούλιο ότι η νομοθεσία στα θέματα αυτά τα δικονομικά είχε καθυστερήσει πολύ. Δεύτερον, δουλεύουμε όσο αποτελεσματικότερα και ταχύτερα γίνεται για να εγκριθούν όλα τα μέτρα. Πέντε είναι στον οδικό χάρτη. Ε, το πέμπτο είναι αυτό το περί και μετάφρασης. Ε, ελπίζομαι η Κομισιόν ε, ε, προβάλλει και τα άλλα, β με ε, πρώτην. Και αρχίζοντας τον Ιούλιο 2010 και θα προχωρούμε με τη σειρά για την ε, υλοποίηση. Μέχρι τον Ιούλιο 2013 με ρυθμό ένα μέτρο κάθε χρόνο. Τρίτον, για το μέτρο Α, η Κομισιόν ήθελε να το προβάλλει αυτό ως σχέδιο οδηγίας, αλλά για θεσμικούς λόγους που εμέσως ανέφερε και ο εισηγητής, δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε τόσο γρήγορα όσο τα κράτη-μέλη που ανακύκλωσαν το κείμενο που συμφωνήθηκε στις 23 Οκτωβρίου για την πρωτοβουλία αυτή. Τέταρτον, το κείμενο αυτό που συμφωνήθηκε στις 23 Οκτωβρίου δέχεται την προσέγγιση του ελάχιστου κοινού παρονομαστή, ενώ τώρα στα πλαίσια της Λισαβόνας δεν το θέλουμε πια αυτό, θέλουμε ε, υψηλότερα στάνταρ στο κείμενο. Θεωρούμε ότι ίσως θα ήταν πιο καλό και πιο σόφρο να επιστρέψουμε στην πρώτη πρόταση του Ιουλίου της Κομισιόν. Γιατί τα πρότυπα και τα στάνταρ προστασίας των κατηγορουμένων είναι υψηλότερα εκεί σίγουρα ως προς ένα-δύο θέματα, ίσως και άλλα. Και ε, ελπίζω σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο να ανεβάσουμε λίγο τα στάνταρ, ώστε το τελικό κείμενο να θυμίζει την αρχική πρόταση της Κομισιόν κάπως περισσότερο. Τέλος, πέμπτη παρατήρησή μου, αυτό το κείμενο, ό,τι και αν εγκρίνομαι θα πρέπει να συνάδει με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η αρχική πρόταση της Κομισιόν του Ιουλίου του 2009 εστάλει στο Στρασβούργο του ώστε οι ειδικοί για τα ανθρώπινα δικαιώματα να το εξετάσουν το κείμενο και να δουν αν ε, είναι εντάξει σε σχέση με τα πρότυπα του Στρασβούργου και δεν θα το σε σχέση με τη σύμβαση. Και θεωρούμε ότι είναι σημαντικό ότι το κείμενο που συζητούμε τώρα να έχει την ίδια σφραγίδα, αν θέλετε, έγκριση από το Στρασβούργο. Γιατί ανησυχούμε λίγο ότι σε κάνα δύο σημεία μπορεί να μην είναι αυτό που πρέπει και να μην συνάδει όπως πρέπει με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Η κυρία Ρωμέρο Λόπες έχει το λόγο. Και εγώ να τονίσω τη σημασία που έχει το γεγονό ότι για την πρώτη πρόταση με, με το νέο θεσμικό πλαίσιο όταν το Κοινοβούλιο πλέον έχει εξουσία λήψης ε, συναπόφασης στον τομέα αυτό και ότι 13 χώρες θεώρησαν αρκετά σημαντικό ένα τέτοιο ζήτημα. Πρόκειται για σημαντικό ζήτημα στα πλαίσια της αναγνώρισης, της ανα, αναγνώρισης των αποφάσεων και της δημιουργία τη αναγκαίας αμοιβαία εμπιστοσύνη που χρειάζεται για να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό δικαστικό χώρο. Στο πλαίσιο αυτό πιστεύουμε ότι το κείμενο καθ' όλη την πορεία μπορεί να βελτιωθεί. Πρέπει να δούμε επίσης και τι σημαίνει η ποιότητα στη διαμηνία και τη μετάφραση και εκεί μπορούμε να προχωρήσουμε περαιτέρω. Πρέπει να σας πω ωστόσο ότι θα πρέπει στο μέλλον να εξετάσουμε κατά πόσο η προθεσμία που προτείνει η Επιτροπή για τα υπόλοιπα δικαιώματα που δεν καλύπτονται εδώ, μια ναι, και μιλάμε για το πρώτο βήμα του οδικού χάρτη και υπάρχουν μια σειρά δικαιωμάτων που δεν υπάρχουν ακόμα και τα οποία η Κομισιόν προτείνει την προθεσμία του ενός έτους για τα υπόλοιπα δικαιώματα. Θα πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσο είναι οι προθεσμίες αυτές, είναι υποχρεωτικές ή κατά πόσο θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε στη δημιουργία του πακέτου το στην ολοκλήρωση του πακέτου αυτού το συντομότερο δυνατό. Μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για ένα χάρτη δικαιωμάτων που εμπεριέχει όχι μόνο τα δικαιώματα των υπόπτων στην ε, διερμηνία και τη μετάφραση, αλλά και την, ε, τα δικαιώματα στην νομική προστασία και ότι η κατάσταση από χώρα σε χώρα είναι τελείως διαφορετική. Υπάρχουν χώρες όπου ε, δεν αναγνωρίζεται το δικαίωμα του κατηγορούμενου στην ε, σιωπή. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να υπάρξουν κάποια κοινά στάνταρ και είναι σημαντικό το πρώτο αυτό βήμα να μην είναι μόνο πρώτο βήμα, να, προχω... τα υπόλοιπα γρήγορα. Γι' αυτό θέλω να ρωτήσω την Επιτροπή σε τι βασίζεται για να θέσει αυτή την προθεσμία του ενός έτους. Δηλαδή πώς μπορεί να προχωρήσει γρήγορα για την υλοποίηση των υπόλοιπων δικαιω, δικαιωμάτων που δεν αναφέρονται εδώ. Πριν την παρέμβαση τη κυρία Λούλινγκ έγινε λόγος, έγινε, τέθηκε το ερώτημα της ε, ε, στη νομική υπηρεσία. Δεν ξέρω αν ε, θέλετε να μιλήσετε. Πάντως, αν γίνει να μιλήσετε σύντομα και να μας βοηθήσετε, θα ήταν χρήσιμο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για τις προσπάθειές σας. Να σας πω, ωστόσο, ότι η κυρία Λάντφορντ με πιάνει τελείως διάβαστο. Προτιμώ να καταλάβω κάπως καλύτερα την κατάσταση, γιατί μία γραπτή απάντηση του Συμβουλίου μπορεί να εξυπηρετήσει και τη σχέση μεταξύ Συμβουλίου και Επιτροπής. Ε, πραγματικά ζητώ την κατανόησή σας γι' αυτό, όχι μόνο τη, ε, τη δική μου και όλων. Είναι γεγονός ότι το κείμενο είναι περίπλοκο και απαιτεί περαιτέρω μελέτη. Κύριε Λάτφορντ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη που ταλαιπωρώ την νομική υπηρεσία. Ίσως ε, καλό είναι να μας απαντήσουν γραπτός. Αν γίνει και έγκαιρα αυτό, πολύ θα το εκτιμήσουμε. Χαίρομαι για τα όσα είπε η Κάρολεν Μόργαν από την Κομισιόν που δούλεψε επί μακρόν για το, πάνω σε αυτό το θέμα. η ηρωίδα είναι. ελπίζω να μην την κάνω να κοκκινήσει. Πρωτοπόρος. Γιατί είναι καλό ότι εγκρίνουμε τον οδικό χάρτη και ένα νομικό μέτρο για τα θέματα αυτά της οικονομίας και ότι θα εγκριθεί από το Συμβούλιο ένα πρόγραμμα δικαιωμάτων για ανθρώπους που βρίσκονται ε, αντιμέτωποι με ποινικέ ε, διαδικασίες. Τώρα, μια πρόταση το χρόνο. Ε, ταχύς ρυθμός είναι για τις Βρυξέλλες. Συμφωνώ με την κυρία Ρομέρο Λόπες όμως ότι όσο πιο γρήγορα τα καταφέρουμε τόσο το καλύτερο. Γιατί δεν θέλουμε... Ε, εδώ, ε, μετά το ευρωπαϊκό ε, ένταλμα σύλληψη εξακολουθεί να υπάρχει ένα μεγάλο κενό και υπάρχουν διαδικασίες που πλέον δεν έχουν νόημα, οπότε χρειάζεται ε, να καλύψουμε το κενό. Πάντως, καλό είναι που ασκούνται πιέσεις υπέρ του μέτρου. Εγώ προσβλέπω στη συνεργασία, όχι μόνο, στενή συνεργασία, όχι μόνο με το Συμβούλιο, αλλά καμιά φορά και με την Κομισιόν, βεβαίω. Γιατί ε, ε, μοιραζόμαστε ε, αυτή τη φιλοδοξία να περάσει αυτό το φιλόδοξο μέτρο. Ωραία. Και γρήγορη και συγκεκριμένη. Να προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο. Περιοριστικά μέτρα καταορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν και το δίκτυο της Αλκάιδα και των Ταλιμπάν. Η συγγήτρια έχει το λόγο, κύριε Μποσκούτ. Θα είμαι πανσύντομη κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι η πρώτη φορά που συζητάμε για αυτό το σημείο, ούτε και τελευταία νομίζω. Θα θυμάστε όλοι αγαπητοί συνάδελφοι, ότι συζητήσαμε πολλές φορές και είχαμε και ένα ψήφισμα εδώ στο Κοινοβούλιο για αυτά τα περιοριστικά μέτρα. Δεν μιλήσαμε μόνο για το περιεχόμενο, μιλήσαμε και για την νομική βάση αυτής της πρότασης ως Κοινοβούλιο και ως Επιτροπή του Κοινοβουλίου είπαμε ότι το άρθρο 75 θα έπρεπε να αποτελεί τη νομική βάση, δηλαδή η συναπόφαση. Αλλά η Κομισιόν και το Συμβούλιο δεν συμφώνησαν μαζί μας. Είπανε ότι το, το άρθρο 215 πρέπει να είναι η βάση και όχι η συναπόφαση. Ζητήσαμε μετά τη γνώμη των νομικών υπηρεσιών του Κοινοβουλίου και φάνηκε σαφέστατα ότι όσον αφορά στο σημείο του Μπιν Λάντεν θα έπρεπε να έχουμε ως βάση το άρθρο 75. Υπόθηκε λοιπόν σαφώς και γύρω από αυτό το θέμα ψηφίσαμε στις 16 Δεκεμβρίου. Παρά λοιπόν τη γνώμη του Κοινοβουλίου για τη νομική βάση, είχαμε πει ότι είχαμε απορίες ως προς την πρόσταση της Κομισιόν και του Συμβουλίου στις 22 Δεκεμβρίου, ελήφθη μία απόφαση σχετικά με τον κανονισμό του Συμβουλίου 1286 του 2009 βάσει του άρθρου 215. Ή, σας είπα ποια είναι η γνώμη του Κοινοβουλίου. Πρέπει να ζητήσουμε λοιπόν την γνώμη του δικαστηρίου για το αρθ βάση του άρθρου 263. Η νομική επιτροπή μπορεί του Κοινοβουλίου μπορεί να συστήσει στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου σχετικά για να προχωρήσει και παρακαλώ την Επιτροπή μας να το υποστηρίξει. Έχετε αντιρρήσεις ε, για την πρόταση της κυρίας Μποσκούχ. Ωραία. Θα προτείνουμε στη νομική επιτροπή τα σχετικά. Τελευταίο σημείο. Ενιαία διαδικασία για άδεια παραμονής και εργασίας. Ο κύριος Μποσουτήλ λοιπόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω ετοιμαστεί για το θέμα, αν και έχω διαβάσει κάποια βασικά ε, σημειώματα. Ούτε η κυρία Μακιό μου είπε ότι δεν θα ερχόταν. Σπάντων, σήμερα αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε είναι να ζητήσουμε το Συμβούλιο κάποιε πληροφορίε σχετικά με την κατάσταση πραγμάτων και την πορεία τη πρόταση. Οπότε, όπως και άλλοι συναδελφοί, θέλω να μας πει το Συμβούλιο όπως έχουν τα πράγματα. Ευχαριστώ. Το Συμβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να σας πληροφορήσω πολύ σύντομα πού βρίσκεται η κατάσταση για αυτό το θέμα που γνωρίζετε όλοι σας πολύ καλά διότι το εξέτασε πολλές φορές το θέμα του Κοινοβούλιο και μπορεί να αποτελέσει και το θεμέλιο για την βελτίωση της κατάστασης των εργαζομένων στην και των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2007 παρουσίασε η Κομισιόν μία πρόταση που τη διαπραγματευθήκαμε στο Συμβούλιο κατά τη Σλοβενική και τη, Γαλλική και τη Τσεχική Προεδρία και το Συμβούλιο δεν καταφέρνει να συμφωνήσει. διότι πρόκειται για ένα κείμενο που, πρόκειται για ένα κείμενο που πρέπει να εγκριθεί ομόφωνα. Είναι αδύνατον λοιπόν να καταλήξουμε σε μία συμφωνία γύρω από αυτό το κείμενο. Υπήρξαν δύο διαφορετικές ε, τάσεις και ευαισθησίες ε, γύρω από αυτό το κείμενο. Ορισμένες χώρες ε, θεωρούσαν ότι το single permit θα έπρεπε να αποτελεί τη λιδία ή λίθο των δικαιωμάτων του κάθε εργαζόμενου που έρχεται εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως όταν έχουμε εγκρίνει άλλες οδηγίες που αφορούν στο θέμα της μετανάστευσης και επίσης ε, είχαμε και, και έπρεπε να εγκρίνουμε μία οδηγία η οποία θα έλεγε ότι όλοι οι μετανάστες εργαζόμενοι που έρχονται στην Ένωση θα πρέπει να έχουν παντού τα ίδια δικαιώματα. Η Τσεχική Προεδρία όμως έλεγε ότι θα έπρεπε να περιοριστούμε μόνο σε διαδικαστικά θέματα που αφορούν σε μία ενιαία άδεια παραμονής ε, και άδεια εργασίας, χωρίς όμως να γίνεται αναφορά στα δικαιώματα αυτής της άδειας. Τώρα με τη Λισαβόνα αλλάζει ριζικά η κατάσταση, το Κοινοβούλιο θα παίξει πολύ πιο σημαντικό ρόλο μέσα από τη συναπόφαση και στο Συμβούλιο τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα γιατί αυτά τα ζητήματα πλέον περνάνε με ειδική πλειοψηφία. Η Κομισιόν έχει καταθέσει το κείμενό της του 2007 στο Κοινοβούλιο και βάσει αυτού του κειμένου θα πρέπει να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Από την Ισπανική Προεδρία θα ήθελα να σας πω ότι για μας το θέμα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό το ξέρει πολύ καλά και η Επιτροπή Λίμπε, θεωρούμε ότι είναι ένα κείμενο το οποίο μετά από το πρόγραμμα της Στοκχόλμης θα πρέπει να προχωρήσει και πριν προχωρήσουμε στη διαπραγμάτευση άλλων οδηγιών πρέπει να ολοκληρώνουμε με αυτό το θέμα. Ε, δηλαδή πριν αρχίσουμε να εξετάζουμε θέματα για τους εποχιακούς εργαζόμενους κλπ. Θα κάνει ό,τι μπορεί η Προεδρία για να προχωρήσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και να συνεργαστεί με τον καλύτερο τρόπο με την Επιτροπή σας και με το Κοινοβούλιο. Η Κομισιόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν έχω να προσθέσω πολλά σε αυτά που είπε η Προεδρία. Απλά να υπενθυμίσω ότι το 7 είχαμε υποβάλει μια πρόταση αρκετά φιλόδοξη. Κάποιοι εδώ την θυμάστε. Είχε πάρει μια πρώτη γνωμοδότηση, το ανέφερε και η Προεδρία. Δεν καταφέραμε ωστόσο να πετύχουμε ομοφωνία στο Συμβούλιο. Τώρα υπάρχει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που να προσθέσω κάτι νομικά ότι το άρθρο 73 της συνθήκης είναι πιο λεπτομεριακό σε διαφορα αφορά τα δικαιώματα των μεταναστών νομίμων κατοίκων της Ένωσης, κάτι που σημαίνει ότι οι εκφράσεις ανησυχία ε, στο Συμβούλιο δεν έχουν πια λόγο ύπαρξης και η νομική βάση του άρθρου 79 διορθώνει ομιλήτρια, επιτρέπει να υπάρξει ευκολότερα συμφωνία για τα δικαιώματα των υπηκών των χωρών. Είναι σημαντική η πρόταση όπως αναφέρθηκε. Υπάρχει μία, είναι μία πρόταση πλαίσιο με πολλά δικαιώματα αφορά ε, απλοποίηση διαδικασιών, ενιαία θηρίδα, ενιαία άδεια παραμονής και εργασίες και πολλά δικαιώματα που είναι πολλά στην πρώτη της Επιτροπής γιατί εμεί προτείνουμε συνθήκες εργασίας μεταξύ των οποίων μισθή, αναγνώριση διπλωμάτων, άδειε κλπ. Ε, πολύ θετικά στο μέτρο που οι εργαζόμενοι από τρίτες χώρες έχουν ίση αντιμετώπιση με τους ημεδαπούς εργαζόμενους. Στο πλαίσιο αυτό το πρόγραμμα της Στοκόλμης τονίζει την ανάγκη να υπάρξει ε, δίκαιη αντιμετώπιση των εργαζομένων. Έχουμε λοιπόν νέο νομικό, νέο θεσμικό και νέο πολιτικό πλαίσιο με το πρόγραμμα της Στοκόλμης που νομίζω ότι θα δώσουν μια νέα όθηση στην, νέα, στην πρόταση αυτή. Όπως αναφέρθηκε, συμφωνίες στο Συμβούλιο το κείμενο τη Συμφωνία του Συμβουλίου ήταν λιγότερο φιλόδοξο από αυτό που σκεφτόταν η Επιτροπή, γιατί το πεδίο εφαρμογή, για παράδειγμα, είχε περιοριστεί μόνο στου κατόχου τη ενιαίας άδεια. Η Επιτροπή πάντα τόνισε ότι δεν μπορούσε να δεχθεί τον περιορισμό αυτό. Η θέση μα παραμένει η αρχική. Θέλουμε να υπάρξει μια φιλόδοξη οδηγία με δίκαιη αντιμετώπιση των μεταναστών και να μην υπάρχουν περιορισμοί μόνο στους ε, κατόχους ενίων αδειών. Όπως επίσης αναφέρθηκε, επιβεβαιώσαμε την θέση μας όταν πέρασαμε στη νέα συνθήκη. Μόνο η νομική βάση και η διαδικασία αλλάζει και δεν είμαστε και είμαστε έτοιμοι συγγνώμη, να συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή για να υπάρξει μια γρήγορη συμφωνία για το κείμενο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. για την ακρίβεια και τη συντομία σε αυτά τα θέματα που είναι ιδιαίτερα ακριβή και σημαντικά. Αύριο λοιπόν θα συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.